Να ξεκινήσουμε το σημείο 8, αγαπητοί συνάδελφοι, που είναι μια παρουσίαση από θεματικό τμήμα για το πολιτική συνοχή. Ουσιαστικά παρουσίαση του θεματικού αυτού τμήματος. Το 60% των βουλευτών είναι καινούργοι, ε, εκλεγέντες και τα θεματικά τμήματα παρέχουν εξαιρετικές ε, υπηρεσίες που δεν τις εκμεταλλευόμαστε. Για να ακούσουμε λοιπόν τι κάνει αυτό το τμήμα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με την ευκαιρία να σας εξηγήσω εν συντομία τι κάνουμε εμείς. Ιδίω ε, σε σχέση και με τη νέα περίοδο αυτή που ξεκινάει το πολιτικό, τα πολιτικά τμήματα δημιουργήθηκαν το 2004 για να στηρίξουν το έργο των επιτροπών και των γραμματιών στο τομέα της έρευνας και της ε, εμπειρογνωμοσύνης. Υπάρχουν θεματικά τμήματα ε, που πλαισιώνουν όλες οι επιτροπές. Όπως βλέπετε καλύπτουμε τις μεταφορές, περιφερειακή πολιτική, την αλία, τη γεωργία, τον πολιτισμό. Όπως είπα, προσπαθούμε να παρέχουμε έρευνα προσανατολισμένη στη δράση παρέχουμε γνωμοσύνη και ε, έρευνα για όλες, ε, για το σύνολο της Επιτροπής, το σύνολο των Επιτροπών και αυτό είναι σημαντικό. Αν κάποιος βουλευτής έχει ένα ατομικό ε, αίτημα και θέλει μια ατομική απάντηση, υπάρχει υπηρεσία έρευνα του Κοινοβουλίου για τα μέλη. Εμεί ε, προσπαθούμε να παρέχουμε στι ανάγκες των επιτροπών ε, υπηρεσίε. Θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο αυτό για να λάβετε τι αποφάσει σα, ε, οπότε προσπαθούμε παραδείγματο χάρη να διευκρινίσουμε τεχνικά, οικονομικά, νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χάραξη πολιτική ή βοηθούμε στην αξιολόγηση της μεταφορά αστικού δίκαιου, τη επιβολή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Πώς το κάνουμε αυτό. Έχουμε δικό μας προϋπολογισμό και σε σχέση με την ερευνητική κοινότητα με την οποία έχουμε άλλη επίδραση. Η εμπειρογνωμοσύνη μας, όπως είπα, προσανατολίζεται στη δράση, είναι action oriented. Προσπαθούμε δηλαδή να δώσουμε κάποιες επιλογές, κάποια σενάρια πολιτικής, τα οποία πιστεύω θα είναι χρήσιμα για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Και προσπαθούμε να αντικαθεπίζονται οι στατηγικές σας προτεραιότητες σε αυτές. Ε, βέβαια, ασχολούμαστε κάποιες φορές με πολιτικά λεπτά ζητήματα. Εστιάζουμε λοιπόν στην αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία. Έχουμε μια σειρά μέτρων ώστε να ε, ισχύουν αυτά που είπα. Έχουμε διαδικασίες προκήρυξης αγωνισμών, πολύ αυστηρά πρότυπα και εντολή. Επιλέγουμε τους εργολάβους με ανταγωνιστική διαδικασία. ένα υπάλληλο του Κοινοβουλίου που πρέπει να έχει και ουδέτερη αμερόληπτη στάση αναλαμβάνει την επιλογή. Έχουμε τη, το peer review και μέτρα κατά της ε, κλοπής, λογοκλοπής και ε, βέβαια θέλουμε να είστε εσείς πιο πολύ ικανοποιημένοι. Ποιες είναι οι μορφές των εγγράφων σύντομα δισέλιδα, τα briefings, ε, αναλύσεις σε βάθος ε, ή μελέτες πάνω από 36 σελίδες. Όλες αυτές οι μελέτες ε, συντάσσονται στα αγγλικά και δημοσιεύονται μόνο στα αγγλικά. Και αυτό για ποιο λόγο, διότι υπάρχουν περιορισμοί στις μεταφραστικές υπηρεσίες που εστιάζουν στο νομοθετικό έργο. Αν υπάρχει όμως συγκεκριμένο ενδιαφέρον για κάποια συγκεκριμένη μελέτη, τότε προσφέρονται καμιά δυο-τρεις άλλες γλώσσες. Αν δεν μπορούμε, ε, αλλά δεν μπορούμε να καλύψουμε τις 24 ε, γλώσσες για τέτοιου είδους μελέτες. Οργανώζουμε επίσης εργαστήρια, διάφορε πάνελ πυρογνωμόνων και άλλες συναντήσεις. Τα έγγραφά μας τα παράγουμε είτε εντός κοινοβουλίου, συνάδελφοι δηλαδή από το θεματικό που είναι ένας μόνο, ο διπλανός μου, αυτή τη στιγμή, λόγω φυσικών περιορισμών. Αλλιώς γίνεται εξωτερική ανάθεση με διαγωνισμό. Και έτσι ερχόμαστε σε επαφή με την ε, κοινότητα των επαϊόντων. Αυτές οι διαδικασίες έχουν ένα μειονέκτημα που είναι διάρκεια. Βλέπετε τι γίνεται. Ξεκινάμε με απόφαση των συντονιστών να γίνει μια μελέτη. Έπειτα. Προκυρίστε τη διακασία διαγωνισμού. Δύο με έξι μήνες διαρκεί η έρευνα. Έπειτα πρέπει να εξασφαλίσουμε τον ποιητικό έλεγχο και αν χρειάζεται ή αν είναι δυνατόν να μεταφραστεί μελέτη, που σημαίνει ότι από την απόφαση των συντονιστών μέχρι την παρουσίαση του εγγράφου μιλάμε για ένα διάστημα από 4 ε, έως 12 μήνες. Αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη σας. Αν για παράδειγμα θέλετε μια συγκεκριμένη μελέτη πριν από μια έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας να έχετε υπολογίσει το χρόνο. Όλα τα κείμενα μας είναι δημοσία προσβάσιμα και από τους συμπολίτες μας ε, μέσω του διαδικτύου. Έχουμε και το ίντρανετ, βλέπετε την σελίδα μας, έχουμε την σελίδα της Επιτροπής ΠΕΧ, το blog, το Twitter και βέβαια υπάρχει και η ε, δυνατότητα να τα συμβουλευτείτε στον τρίτο όροφο του ΑΣΠΑ και στη βιβλιοθήκη αυτά τα έγγραφα. Να πω σύντομα δύο λόγια για το τι κάναμε στην τελευταία θητεία και τι προβλέπετε να συντάξουμε στην προηγούμενη Επιτροπή ΠΕΣ είχαμε 42 εξωτερικές μελέτες για τη διαχείριση των ελευμάτων, την Αρκτική, στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, για τα παρασυρώμενα πλάδια, για την εκπαίδευση. Είχαμε επίσης ε, workshop για την ε, κοινή πολιτική, βιώσιμη ανάπτυξη, μπλε Brexit και πολλά άλλα. Ποιε είναι οι δύο μελέτε που αναμένεται να σα παρουσιάσουμε. Η μία είναι οι τελευταίε εξελίξει και μελικέ προκλήσει για την αλληλευτική πολιτική και η άλλη είναι η βιομηχανία των θαλασσινών και πώς αυτή ενσωματώνεται στην Ένωση και τα κράτη-μέλη που έχουν ακτογραμμή. Για το σχεδιασμό τώρα που ξεκινάμε θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με εσά για να μας δώσετε τις ιδέες σας για το τι θα θέλατε να εκπονήσουμε για το πρώτο εξάμεινο του 2020. Βράτω με δε της ευκαιρίας για να τονίσω πως για μας είναι πολύ σημαντικό το feedback από εσάς, γιατί έτσι θα είμαστε και εμείς βέβαιοι ότι παράγουμε ε, έργο το οποίο εσείς χρειάζεστε. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Δύο τουλάχιστον συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Να πω ότι θυμάμαι το κοινοβούλιο του 99 Και είναι σημαντικό ότι αφαιρώσαμε τόσου πόρου στην έρευνα για να μπορούμε να λέμε κάποια πράγματα με το σχετικό κύρος. Για τα μέλη μα, αν έχετε ιδέε για θέματα προ ε, διερεύνηση, πείτε το στους συντονιστές σας, διότι μπορούν να το θέσουν σε κάποια συνεδρίαση, να το, να το συζητήσουμε ε, εντάχει και να προωθηθεί προ τι αρμόδιες υπηρεσίες για να παραγγείλουμε κάποια έρευνα. Όποιο λοιπόν έχει κάποια ιδέα, κάποια παρατήρηση, κάποια ομάδα έχει κάτι να πει, ε, είμαστε στη διαθέσή σα. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε σε ένα παράδειγμα τη δουλειά σα. Η προηγούμενη Επιτροπή παρήγγειλε μια μελέτη για τις τελευταίες εξελίξεις και τις μελλοντικέ προκλήσεις για την αλληλευτική πολιτική. Και ε, η μελέτη αυτή διεξήχθη από τρία μεγάλα ιδρύματα. Το Πανεπιστήμιο της Βρετάνης της Γαλλίας, το Πανεπιστήμιο Νομίζω τώρα μοιράζεται η έκθεση και επίσης από το Πανεπιστήμιο Άκουα της Δανίας και το Άστι Τεκνάλια της ε, Ισπανίας. Θα δούμε λοιπόν εδώ πέρα την ε, κοινή οργάνωση αγορών και την εξωτερική διάσταση. Θα ζητήσω από τον ε, καθηγητή Λεγκαλίκ της Δυτικής Βρετάνης να μας παρουσιάσει τα θέματα της ΚΟΑ, της κοινή οργάνωσης αγοράς. Κύριε Λεγκαλίκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω την παρουσίασή μου θυμίζοντας το γενικό στόχο της μελέτης αυτής να δώσουμε μια συνολική επισκόπηση στην Επιτροπή Αλίας του Κοινοβουλίου για τα στοιχεία που προέκυψαν σε διαφορετικούς τομείς της αλίας κατά τη διάρκεια προηγούμενων θητιών και να εντοπίσουμε αυτά που θεωρήσαμε βασικά προβλήματα, βασικές προκλήσεις. Αυτά που θα σας παρουσιαστούν σε ένα προσεχές ή ιδιαίτερα προσεχές μέλλον. Αυτά που θέλω εγώ να σας παρουσιάσω έχουν να κάνουν με τις κοινέ οργανώσεις αγορών, της ΚΟΑ. Και θα διερθώσω την παρουσίασή μου ως εξής. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω υπενθυμίζοντας τους στόχους της κοινή οργάνωσης αγορών. Μετά θα παρουσιάσω τέσσερις, τέσσερα στοιχεία που έχουν θεωρηθεί ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ενδιαφερουσών προσφάτων εξελίξεων μετά θα απαριθμίσω μια σειρά από μελλοντικέ προκλήσεις, οι οποίες αναλύονται λεπτομερώς στην έκθεση και εδώ θα φανούν ξεκάθαρα μέσα από τρία case study, μέσα από τρεις συγκεκριμένε υποθέσεις που μελετώνται, ώστε να δούμε τις κατηγορίες προκλήσεων που μπορεί να έχουμε να αντιμετωπίσουμε και στο, και στο τέταρτο σημείο θα αναπτύξω κάποια συμπεράσματα. Καταρχάς, για τους στόχους της κοινή οργάνωσης αγορών. Εάν ο γενικός στόχος αυτού του νομοθετήματος είναι να διευκολύνει την επίτευξη των στόχων της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, είναι ξεκάθαρο ότι οι ΚΟΑ σκοπό έχουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τις οικονομικές επιδόσεις των παραγωγών κατά τρόπον ώστε να τις διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα και να αποκομίσουμε τα υψηλότερα δυνατά οικονομικά ωφέλη. Αυτό βασίζεται σε κάποιες προϋποθέσεις, κυρίως τη σταθεροποίηση των αγορών. Το γεγονός ότι η ανταγωνιστικότητα είναι όσο το δυνατόν υγιέστερη μεταξύ Ευρωπαίων και έξω Ευρωπαϊκών παραγωγών είναι ένα καθοριστικό στοιχείο. Επίσης θέλουμε να προωθήσουμε την πλέον ποικίλη προσφορά ε, προϊόντων θαλάσσιων από την, προς τον καταναλωτή, ιδίως θαλάσσιων προϊόντων από τα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς τις πρόσφατες εξελίξεις πρέπει να θυμίσω κάποια στοιχεία που προέρχονται από την τελευταία έκθεση του CSTP. Ε, δείχνουν ότι τα προηγούμενα χρόνια οι οικονομικές επιδόσεις ως προς την αλία έχουν αυξηθεί σήμερα. Φτάνουμε μια ακαθάριστη γενική αξία που ξεπερνάει τα 85 εκατομμύρια ευρώ και την ε, αξία να φτάνει τα 2 δις. Αυτό έχει να κάνει με συγκεκριμένα στοιχεία, στοιχεία διαρθρωτικά, τα οποία σε κάποιο βαθμό οδήγησαν σε μείωση των ελευθερικών δυνατοτήτων Θα αφήσω την ε, συνάδελφο να τα αναπτύξει. Έπειτα είχαμε καλύτερη διαχείριση των αλληλευτικών δυνατοτήτων από την πλευρά ιδίω των οργανισμών διαχείρισης και των, οργανισμών των, παραγω... των οργανώσεων των παραγωγών. Άλλα στοιχεία που έχουν θεωρηθεί καθοριστικά και από τους εκπροσώπους της, της αλληλευτικής βιομηχανίας αλλά και από τους αναλυτές είναι η σταδιακή θέσπιση νομοθεσίας. Νομοθεσίας που σκοπό έχει να αντιμετωπίσει τα προϊόντα της λεγόμενης παράνομης, άναρχης και άτυπης αλίας προκειμένου να διασφαλίσουμε την ίση μεταχείριση των Ευρωπαίων παραγωγών. Ιδίως σε συγκεκριμένα ε, τμήματα της αγοράς. Εδώ να θυμίσω ένα γεγονός που συχνά το ξεχνάμε, αλλά που η νέα νομοθεσία το έλαβε υπόψη. Χρειάζεται χρόνος Και ακόμη και αν η νομοθεσία αυτή εγκρίθηκε το 2008, χρειάστηκαν χρόνια και χρόνια για μια καλή εφαρμογή της. Ένα άλλο στοιχείο που είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι πραγματικά ορόσημο αλλαγή της νοοτροπίες είναι η πάυση δραστηριότητα. Δηλαδή, οι αλλοί μπορούν να πάρουν αποζημίωση όταν δεν βρίσκουν αγοραστή και τα ψάρια πρόκειται να απομακρυνθούν ω απόρριμα. Αυτό από περιβαλλοντική άποψη και από οικονομική σκοπιά μπορεί να ήταν ιδιαίτερα επωφελέ και για κάποια χρόνια ήταν φαίνεται αδύνατο να καταργηθεί. Όμως τελικά ο μηχανισμός αυτός καταργήθηκε χωρίς να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα εκτός από τους πρώτους μήνες της εφαρμογής. Τέλος και πάντοτε σε σχέση με τις ανησυχίες στις ίδιες τις αγορές για τη γενική διαδικασία διαχείρισης της αλίας, κατά την προηγούμενη θητεία εγκρίθηκε αυτό που ονομάζουμε προγράμματα εμπορίας, παραγωγής και εμπορίας. Αυτό υποχρεώνει κάθε οργάνωση παραγωγών να προβλέψουν στα προγράμματα παραγωγής τους και στα προγράμματα διαχείρισης τις ανησυχίες της αγοράς. Και αυτό αναπτύχθηκε δραστικά τα τελευταία χρόνια. Ένα άλλο σημείο που δεν θέλω να το θίξω εδώ ήταν η εξέλιξη των δυνατοτήτων. Δυνατοτήτων ανάλυσης των δεδομένων με την σταδιακή ανάπτυξη εργαλείων όπως το παρατηρητηρίο των αγορών, το ΕΜΟΦΑ, για να καταλαβαίνουμε καλύτερα τα θέματα που προκύπτουν. Τώρα θα περάσω σε κάτι που για σας ίσως να είναι σημαντικότερο. Διότι αρκετά γρήγορα θα πρέπει να ασχοληθείτε με το θέμα. Οι βασικές μελλοντικέ προκλήσεις. Στην έκθεση απαριθμώνται κάποιες μελλοντικέ δυσκολίες και εδώ θέλω να παρουσιάσω τριών ειδών προκλήσεις, τρεις κατηγορίες και η κάθε μια βασίζεται στη μελέτη μιας συγκεκριμένη υπόθεσης, μιας περίπτωσης που μπορείτε να βρείτε και στην έκθεση. Η πρώτη είναι να διασφαλίσουμε την ε, ισότιμη η αποτελεσματική ανταγωνιστικότητα μεταξύ παραγωγών mm. και όλος ιδιαίτερος μεταξύ των Ευρωπαίων παραγωγών σε αντιδιαστολή με τους εξωευρωπαϊκούς. Αυτό σε ένα πλαίσιο όπου βλέπουμε να υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση όλο ένα και περισσότερε συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών και τελωνιακέ ενώσει. Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι παραγωγοί πολλέ φορέ πρέπει να ανταγωνιστούν απευθεία ε, παραγωγού άλλων περιοχών του κόσμου που δεν υπόκειται στους ίδιους κανόνες, στην ίδια νομοθεσία. Αυτό, μακροπρόθεσμα, μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά προβλήματα. Και αυτό αναφέρεται κυρίως και στο σημείο 4 της, ε, του κανονισμού για τις κοινέ οργανώσεις αγορών λέγεται ότι όταν ενδιαφερόμαστε για διεθνείς συναλλαγές πρέπει παρόλα αυτά να λαμβάνουμε υπόψη το σύνολο των στοιχείων της βιωσιμότητας, της αεφορίας των συστημάτων παραγωγής συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών προδιαγραφών που ισχύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα στοιχείο κλειδί φαίνεται να είναι εδώ ότι το σύνολο των στοιχείων της αηφορία και τη βιωσιμότητα θα πρέπει να μπορούν να ελέγχονται. Και όλα αυτά, για να τα αποδείξω, θα σας πω πολύ γρήγορα μια, τι γίνεται με μια περίπτωση που μελετάτε στην έκθεση, γνωρίζοντας όμως ότι είναι ένα παράδειγμα μεταξύ άλλων. Πρόκειται για την υδατοκαλλιέργεια των ε, ε, για το λαβράκι και την τσιπούρα που έχουμε στην Γαλλία και την Ιταλία. Ε, η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη όμως παραγωγή στην αγορά αυτή τη στιγμή είναι η Τουρκία. Και επειδή στην τελευταία έκθεση του Π τα είδαμε αυτά, Βλέπουμε ότι οι προδιαγραφέ περιβαλλοντική και κοινωνικέ στην Τουρκία δεν είναι οι ίδιε με τι δικέ μα. Οι Τούρκοι παραγωγοί λοιπόν προτείνουν δύο φορέ φτηνότερα προϊόντα από τα δικά μα. Άραγε μπορεί να μην το βλέπετε στη διαφάνεια, είναι μικρή η αριθμή. Έχουμε οικονομικές επιδόσεις που είναι πολύ χαμηλές για το σύνολο του τομέα αυτού και μάλιστα δυναμικό πολύ χαμηλότερο από το σύνολο, από το κανονικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να γνωρίζετε ότι από το 2012 οι Τούρκοι έχουν υποκαταστήσει τους Έλληνες στην αγορά εξαγωγών προς την Ισπανία. Και ένα μέρος αυτής της ε, βιομηχανικής παραγωγής θα πάει κατευθείαν στην Τουρκία. τι μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι η νομοθεσία που προβλέψαμε για να καταπολεμήσουμε την ε, παράνομη, παράτυπη και άναρχη αλία είναι ένα καλό πρωτοβήμα. μπορούν οι νόμοι που θα προβλεφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλουν στο ίδιο επίπεδο ανταγωνισμό όλους τους παραγωγούς. Το σύνολο των στοιχείων που αποτελούν το σύστημα της παραγωγής πρέπει να μπορούν να ελέγχονται, να παρακολουθούνται και να επαληθεύονται. Ιδίως ό,τι αφορά την ε, ε, διατροφή των ζώων των οργανισμών ή αντιβιωτικά που μπορεί να μην επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά επιτρέπονται αλλού. Όλα αυτά τα συστήματα παραγωγή πρέπει να ελέγχονται γιατί μετά όλα αυτά τα στοιχεία νομίμω μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρομοίω, η οδηγία της, ε, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για τις εργασιακές προδιαγραφές θα υλοποιηθεί σε όλες τις χώρες. Όμως, αυτό και πάλι μπορεί να είναι διακριτική μεταχείριση γιατί είναι άλλη νομοθεσία που ισχύει τώρα και άλλο και το κόστος προφανώς. Οπότε δεν γίνονται οι ίδιες κοινωνικές προδιαγραφές παντού σεβαστές με τον ίδιο τρόπο. Ιδίω για τι εξόχω απόκεντρε περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω λέγονται αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Διότι για τα ίδια είδη μπορεί η παραγωγή να, έχουν, να ε, ε, υποβληθούν σε διαφορετικούς κανόνες. Και μετά θέλω να αναφέρω ένα άλλο είδους δυσκολία που έχει να κάνει με το γεγονός ότι σήμερα ένα σημαντικό μέρος των προϊόντων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγονται στόχος της κοινή οργάνωσης αγορών είναι να αντλήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από τους πόρους που διαθέτουμε στα ευρωπαϊκά ύδατα. Το 43% της ευρωπαϊκής παραγωγής βασίζεται σε πέντε είδη. Πέντε είδη τα οποία κυρίως εισάγονται, όπως ο τόνος, ο σολομός, ο μπακαλιάρος της Αλάσκας και οι γαρίδες, κυρίως οι τροπικές γαρίδες. Αυτά έχουν μεγάλη σημασία για βόρειε και βορειοδυτικές χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι κατοχώρες, η Πολωνία, όπου τα πρώτα είδη είναι περίπου το 70% της ε, κατανάλωσης. Αυτό προκύπτει από πολλά φαινόμενα που συνδυάζονται μεταξύ τους. Κυρίως στρατηγική των παραγωγών από τη μία και την ανάγκη να δυσδύσουν σε κάποιες αγορές για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Αυτό συμβαίνει και σε έρκετες ευρωπαϊκές χώρες. Και το άλλο έχει να κάνει με τις γνώσεις των καταναλωτών και τα ίδια τα προϊόντα. Όσο περισσότερα γνωρίζουν και τα εμπορικά προϊόντα, όσο πιο πολύ διαδοθούν τα εμπορικά προϊόντα, τόσο πιο πολύ θα ε, γίνουν για τόσο πιο πολύ θα είναι γνωστά τα προϊόντα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως η όπως για την γενέδος γλώσσας που στην αρχή ήταν πολύ δημοφιλές και μετά περιορίστηκε η κατανάλωσή της. Αυτό μας δείχνει ότι κάποια, κοινοτικά, κάποια είδη που καταναλώνται πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, καταναλώνονται στην Ευρώπη ε, από την τοπική παραγωγή. Τα ετήσια ποσοστά δείχνουν ότι μόνο στην Πορτογαλία ξεπερνάμε τα 300 ευρώ ανά ε, το χρόνο ανά νοικοκυριό. Στι περισσότερε χώρε είμαστε στα 200 ευρώ και λιγότερο. Αν το συγκρίνουμε με την κατανάλωση των προϊόντων με σάρκα σε άλλες χώρες, βλέπουμε ότι είμαστε πολύ κάτω από το μέσο επίπεδο διατροφής. Εδώ πρέπει να βρούμε νέους τρόπους να επικοινωνούμε, ιδίως για τα διατροφικά στοιχεία τα θρεπτικά στοιχεία των προϊόντων της θάλασσας και κυρίως τι γίνεται με τις νέες γενιές που απομακρύνονται από τα παραδοσιακά προϊόντα της θάλασσας. Και πρέπει να πληροφορήσουμε, να ενημερώσουμε για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια διεθνή αλυσίδα παραγωγής προϊόντων της θάλασσας και να ενημερώνουμε για το πώς μπορούν να καταναλωθούν τα επεξεργασμένα προϊόντα. Αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό. Όταν όμως είναι, πρέπει να ενθαρρύνουμε την, την κατάσταση των ε, εισαγόμενων από προϊόντα ευρωπαϊκά. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι τα προϊόντα όπως ο καπνιστός Σολομός. Η Γαλλία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στην κατανάλωση ευρωπαϊκού ε, ε, καπνιστού Σολομού που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αντικατασταθεί από καπνιστή πέστροφα ευρωπαϊκής παραγωγής. Έχουμε και τεχνογνωσία, έχουμε και πόρους, η αγορά υπάρχει. Επίσης, είναι δυνατόν κάποιοι δημόσιοι κρατικοί θεσμοί να παίξουν κάποιο ρόλο προς την ε, ενημέρωση και την εκπαίδευση για τη διατροφή. Μπορούν στα κρατικά εστιατόρια, στις καντίνες, να προωθήσουν μια ε, κατανάλωση τέτοιων προϊόντων. Αυτό μπορεί να γίνει σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση ως προς την κερδοφορία. Τι σημαίνει αυτό. Σήμερα δεν έχουν όλες οι εταιρείες της Ευρώπης καλές οικονομικές επιδόσεις και σε κάποιες περιπτώσεις στις ευρωπαϊκές χώρες έχουμε ελεκτικές δραστηριότητες που μπορεί να βλάψουν άλλες παράλληλες αλληλευτικές δραστηριότητες αλλά ιδιαίτερα κερδοφόρες αυτές με μεγάλη παραγωγή. Αυτό το λέει με λεπτομέρειες κατά λεπτός η έκθεσή μας που δείχνει ότι για μία αλληλευτική δραστηριότητα μπορεί να υπάρχει διαφορετική ανάλυση του κόστους και διαφορετική ανάλυση του, των οικονομικών απολαβών ανά είδος. Αυτό είναι σημαντικό και στα πλαίσια του άρθρου 17 της κοινή αλληλευτικής πολιτικής που ζητά να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια, τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και τα περιβαλλοντικά πρότυπα στην ε, κατανομή των πόρων. Βλέπετε εδώ κάποια παραδείγματα των διαφορών που μπορεί να προκύψουν στις τιμές για το ίδιο είδος. Είτε ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής, είτε ανάλογα με τις διαφορές της χώρες με διαφορετικό τρόπο παραγωγής. Βλέπετε ότι με το λιθρίνι που ψαρεύεται λόγου χάρη με ε, το καλάμι ή με δίχτυ μπορεί να υπάρχει διαφορά στην τιμή. Επίσης βλέπετε διαφορετικά συστήματα ε, παρασυρώμενων δικτυών που ε, αναφέρονται στην έκθεση μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας. Επίσης, μπορούμε να δούμε ότι μεταξύ των διαφορετικών χωρών έχουμε άλλες οικονομικές επιδόσεις λόγω των πόρων. Βλέπετε, ας πούμε, ότι εκεί που είναι πιο αυστηρή η νομοθεσία τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε αύξηση στην παρουσία των αποθεμάτων. Στρέφομαι προς την Κλάρα, αλλά νομίζω δεν είχαμε τόσο υψηλά επίπεδα εδώ και χρόνια. Ενώ εκτός των ζωνών αυτών που υπόκειται σε αυστηρή νομοθεσία, τα αποθέματα αρχίζουν να φθήνουν. Άρα θα μπορούσε να υπάρχει ανάλογη αύξηση στα αποθέματα αν ήταν ανάλογη και η διαχείριση στα, ε, στην αλία. Και τώρα κάποια συμπεράσματα για να περάσω μετά στι συστάσει. Για όσου δουλεύουν, για τα θέματα, δουλεύουν στα θέματα αυτά, για τη διαχείριση τη Αλία εδώ και 20 χρόνια, είναι σαφές ότι έχουν γίνει σοβαρά βήματα πρόοδου σε σχέση με τα τέλη τη δεκαετία του 90. Ωστόσο, Ακόμη υπάρχουν μεγάλα, μεγάλα, μεγάλες περιοχές δραστηριότητας που θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις οικονομικές επιδόσεις από την αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων ή αυτών που των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας. Ε, έχω υπόψη μου εδώ τις εταιρείε αλλά και τους ίδιους τους παραγωγούς. Διότι βλέπουμε ότι το τομέας της αλίας σήμερα σε πολλές χώρες μπορεί να οδηγεί σε πολύ Ενδιαφέρουσε απολαύε. Στην περίπτωση τη αυτοκαλλιέργεια. μπορούν τα πράγματα να πάνε καλύτερα, όμως αυτή τη στιγμή είναι πολλές ε, και αυστηρές είναι πολύ και αυστηροί οι κανόνες που εφαρμόζονται λόγω της νομοθεσίας. Είναι πιο ε, δύσκολο να είναι ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή παραγωγή δηλαδή. Και μετά αναφέρθηκαν και προηγουμένω κάποια στοιχεία. Το γεγονό ότι οι οικονομικές επιδόσεις Κάποιες φορές συνδέονται με το σύστημα διαχείρισης, ιδίως για τα κοινά συστήματα παραγωγής, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ιδίως για το ίδιο είδος, τη στιγμή που αλλιεύεται, μπορεί να πουληθεί σε καλή τιμή, αρκεί να βρεθεί και η σωστή αγορά. Αυτό το έχουμε δει στο παρελθόν για είδη όπως ε, για το και κάποιο καλαμάρι που τελικά βρήκε τον δρόμο του προς την αγορά. Τρεις συστάσεις τώρα. Ε, υπάρχουν χώρες που είναι σημαντικοί, σημαντικές στην αγορά των προϊόντων της θάλασσας. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει υγιής ανταγωνισμός εδώ. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί να αντιμετωπίζουν τις ανάλογες προκλήσεις μάλλον με αυτές των ε, μη Ευρωπαίων Πρέπει να προωθήσουμε τα είδη που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στα ευρωπαϊκά είδατα, αλλά τα υποτιμάμε. Διότι δεν περνάνε από τους σωστούς διάβλους παραγωγής και πρόωθησης, δηλαδή τα μεγάλα σούπερ μάρκετ στην πραγματικότητα. Οι δημόσιες αρχές εδώ μπορούν να παίξουν ένα ρόλο εκπαίδευση σε πρώτη φάση και σίγουρα υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης σε αυτό το επίπεδο. Και ε, τέλος πρέπει να μπορέσουμε στους φορείς διαχείρισης, ιδίως της ΚΟΑ και στα μέλη τους, την δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν σε διαφορετικές αγορές, ιδίως με καλύτερη εκπαίδευση σε θέματα οικονομικής απόδοσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε τον καθηγητή, ε, ο οποίο ζήτησε να είναι πρώτο, γιατί μάλλον επειδή χρειάζεται να αποχωρήσει. Δεν ξέρω αν τα μέλη θα ήθελαν τώρα το λόγο. Παρακαλώ, κυρία Αγγιλέρα. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και ήθελα να ευχαριστήσω, Πρόεδρε, θερμά μας εξηγεί πώς ε, λειτουργεί η ΚΟΑ στα πλαίσια της αλίας. Εγώ εγνώριζα τη ΚΟΑ περισσότερο στα τρόφιμα, τα λοιπά τρόφιμα δηλαδή, και εκτίμησα πολύ την παρουσίαση αυτή. Ήθελα λοιπόν ε, κάποιες ε, διευθυνιστικές ερωτήσεις να κάνω. Από τα όσα είπατε, προκύπτει ότι υπήρξε χρήσιμη εικόα, αλλά υπάρχει και, υπάρχουν κάποιες σημαντικές ελλείψεις. Οι τιμές, αφενός, και ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει επί των προϊόντων αλληλείας η οδηγία που εγκρίναμε πρόσφατα, εδώ και κάποιους μήνες, για τις ε, έκνομες εμπορικές πρακτικές και για προϊόντα αλληλευτικά. Όταν αυτή θα μετεγγραφεί λοιπόν στην νομοθεσία των κρατών μελών, θα μπορούσε αυτό να έχει ένα θετικό αντίκτυπο για τα προϊόντα τα αλλιευτικά και συνολικά τα γεωργικά προϊόντα. Επίσης, τι επιρροή μπορούν να έχουν οι, οι κανόνες ε, της ε, προστατευμένης προέλευσης, της ε, ονομασίας προέλευσης στα προϊόντα τα λιευτικά. Και εδώ δεν ξέρω αν έχουμε λάβει υπόψη μας συνολικά τι δυνατότητες μπορούμε να έχουμε από την ονομασία προέλευση από τις προστατευμένες γεωγραφικές ονομασίες. Η εισαγωγή λοιπόν διεπαγγελματικών συσχετισμών, διακλαδικών συσχετισμών σε όλη την τροφική αλυσίδα και τελικούς μέχρι τον καταναλωτή. αυτά ε, στις κατηγορίες των τροφίμων έχουμε, έχουν τα στοιχεία αυτά τα, της διεπαγγελματικής ε, προσέγγισης πολύ ευεργετικές επιρροές ε, στα γεωργικά προϊόντα, αλλά θα μπορούσαν να έχουν και στα αλλιευτικά. όπου μπορεί ο ένας τομέας να υποστηρίξει τον, τον άλλο. όπως συμβαίνει και στον αλλιευτικό τομέα, τομέα αντίστοιχα ε, ως προς τον αντίκτυπο της παράνομης και λαθρείας αλίας. Όταν συνάπτουμε συμφωνίες με τρίτες χώρες οι οποίες δεν καταπολεμούν αποτελεσματικά την IUU. Έχουμε τέτοιο αντίκτυπο και αν απαιτούσαμε τις ίδιες προϋποθέσεις και από τους εταίρους μας, από τις τρίτες χώρες, θα είχαμε ένα πιο ισότιμο παιχνίδι. Και δίνω εδώ ως παράδειγμα το Βιετνάμ εκτός άλλων χωρών. διάφορα τέτοια στοιχεία και οι διατάξεις της οδηγίας ε, για τον, για τον δίκαιο ανταγωνισμό θα μπορούσαν να έχουν επιρροή σε όλα αυτά. Δηλαδή, λέει ο πρόεδρος, εννοείται μη δασμολογικά εμπόδια. Ε, δεν ξέρω δηλαδή πώς θα μπορούσε να το ερμηνεύσει κανείς αυτό με άλλο τρόπο. Τέλος πάντων, ας ακούσουμε τον επόμενο μιλητή Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον καθηγητή για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση. Εγώ συμφωνώ με την ανησυχία που έχει εκφραστεί για την πολύ χαμηλή διαφάνεια προέλευσης των αλληλευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Δεν βοηθούν όλα αυτά για την αποτελεσματική ενημέρωση του καταναλωτή. Η χαμηλότερη τιμή λοιπόν ενός εισαγόμενου προϊόντος θα μπορούσε να κρύβει πολύ χαμηλή κοινωνική αλλά και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Όλα αυτά ε, την ώρα που εκφράζεται μια πλειοψηφική ικανοποίηση ε, των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα εισαγόμενα προϊόντα και όλα αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο επί του δικού μας κλάδου. Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε μια συγκεκριμένη ε, επισήμανση, ετικετοθεσία, ε, Βιώσιμη αλλιευτική παραγωγής για τα προϊόντα μας και αν θεωρείτε ότι θα μπορούσαν τα αλλιευτικά προϊόντα τρίτων χωρών θα μπορούσαν να υπόκεινται σε ένα σύστημα πιστοποίησης ε, ώστε να βεβαιώνεται η συμμόρφωσή τους προς τα πρότυπα, τα γεωργικά και αλλιευτικά που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε από την προηγούμενη εντολή ένα ε, έργο ευρωπαϊκό που αφορούσε στα, στη διατροφή στα σχολεία. Αυτό θα μπορούσε να τον μιμηθούμε και στα αλληλευτικά προϊόντα, π.χ. όπως είχε ονομαστεί και εκείνο το πρόγραμμα, αυτό να το λέγαμε fish and chips στο σχολείο. Μάλιστα λέει ο Πρόεδρος. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον συντάκτη της έκθεσης Τη μελέτη που μας έκανε και την παρουσίαση, πρώτα απ' όλα κάποια γενικά σχόλια και μετά τρεις σύντομες ερωτήσει. Γενικώ πρώτα. Πριν από μερικά χρόνια όταν άρχισα να εργάζομαι σε αυτή την επιτροπή, αυτές οι μελέτες συνήθω διατίθενταν, διατίθενταν στις ε, διαφορετικές γλώσσες εργασίας στα μέλη τη επιτροπή. Αυτό σταδιακά άλλαξε. Κάθε φορά παίρναμε σε όλο και λιγότερες γλώσσες τις μελέτες και κάποιες φορές μόνο σε μία. Κάποιες φορές ζητάγανε βουλευτές να μεταφραστούν οι μελέτες σε γλώσσες που αρχικά δεν προβλεπόταν. Τώρα βλέπουμε αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει καμία διάθεση επένδυση σε αυτό το εργαλείο που θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο εάν το γνωρίζαμε όλοι και ξέραμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το ότι δεν μεταφράζονται τα κείμενα για του βουλευτέ περιορίζει τη δυνατότητα αντίδρασή μα και την αποτελεσματικότητά μα. Και ε, απευθύνομαι και στου συντονιστέ εδώ. Κύριε Πρόεδρε, κάντε ό,τι μπορείτε εδώ. Ε, ό,τι περνάει από το χέρι σας για να αλλάξει αυτή η τακτική. Και αν γίνεται αυτές οι μελέτες, εάν όχι, τουλάχιστον κάποιες όπως αυτή, να διατίθενται και σε άλλες γλώσσες, στις διάφορες γλώσσες εργασίας μας. Αυτό ήταν το πρώτο σχόλιο και τώρα για τα υπόλοιπα σημεία. Η μελέτη αυτή μου φαίνεται άκρο ενδιαφέρουσα, όχι μόνον επειδή μας επισημαίνει μια νέα πραγματικότητα, αλλά γιατί ακριβώ επιβεβαιώνει σημαντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πραγματικότητα του τομέα της αλίας. Το πρώτο σημείο που βλέπουμε να επιβεβαιώνεται είναι ότι ζούμε σε μια κατάσταση αθέμητου ανταγωνισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα, οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που έχει συνάψει, τελικά βλέπουμε να πλήττει τον τομέα της αλίας που έχει πεσμένους αριθμούς και χειρότερες οικονομικές και κοινωνικές επιδόσεις. Θυσιάζουμε δηλαδή την ε, πολιτική της αλίας στο βωμό ε, των εμπορικών συμφερόντων της Ένωσης που αυτή τη στιγμή προωθούνται και θεωρούνται τα σημαντικότερα. Ιδίως για τα τμήματα του στόλου που είναι τα πιο ευπαθή και σε χώρες που έχουν περισσότερες δυσκολίες και είναι δυναμότερες οικονομικά και κοινωνικά. Το δεύτερο σημείο που θεωρώ σημαντικό από την παρουσίαση που ακούσαμε, διότι ήταν σαφής η μελέτη στα συμπεράσματά της εδώ. Νομίζω η παρουσίαση ήταν πραγματικά εύγλωτη. Έχουμε απέναντί μας μια πραγματική αποτυχία του συστήματος των κοινών οργανώσεων αγορών για τους αλείς. Το είπατε ξεκάθαρα. Ένας από τους βασικούς στόχους των ΚΟΑ που ήταν να διασφαλίσουν την αξιοποίηση Τη της αλλιευτικής δραστηριότητας ή τέλος πάντων τα αλλιεύματα των στόλων των κρατών μελών να φέρνουν ανάλογες απολαβές στους ψαράδες, στους αλλιείς, αυτό απέτυχε. Αυτό θα έπρεπε κάποιο να του οδηγήσει σε σκέψει. Η κατεύθυνση που πήραμε, η οδό που ακολουθούμε, να, να εξαρθρώσουμε σιγά σιγά ε, τι κοινέ οργανώσει αγορών, τα εργαλεία ε, ρύθμισης που υπήρχαν δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Μεγαλύτερη απελευθερώση του τομέα της αλίας ε, τελικά ήταν αυτό που προκρίναμε. Δεν πετύχαμε καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων και περισσότερες απολαβές για τους αλείς. Αυτό θα πρέπει ε, να οδηγήσει σε σκέψεις ε, αυτούς που άνοιξαν το δρόμο στην απελευθέρωση για το τι τελικά πετύχαμε. Τι πετύχαμε. Μια ευκαιρία για μεταρρύθμιση της αλληλευτικής πολιτικής που μάλλον θα πρέπει να μας οδηγήσει σε ενίσχυση των προηγούμενων εργαλείων ρύθμισης για να μπορέσουμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε αυτά που έχουμε αλλιεύσει, τα αλλιεύματα και να φέρουμε δίκαιες απολαβές στους ε, ψαράδες. Και κάτι ακόμα που θεωρώ σημαντικό από την παρουσίαση που ακούσαμε, οι διαφορετικές ε, κερδοφορίες, για να τις πω έτσι, του τομέα αυτού έχουν να κάνουν και με το κάθε τμήμα του στόλου για το οποίο συζητάμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί κάποιε φορέ εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μα λέει ότι η κοινή ελευθερική πολιτική ήταν επιτυχία. Διότι η κερδοφορία του τομέα αυξήθηκε τόσο τα τελευταία τάδε χρόνια. Η μελέτη όμω αυτή δείχνει και επιβεβαιώνει την πραγματικότητα ότι υπάρχουν διαφορετικέ καταστάσει σε κάποια κρατημέλη. Κάποιοι αυξήσαν τα κέρδη του και κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιοι τα πήγαν καλά και άλλοι τα πάνε πολύ άσχημα για να μην πω και πολύ άσχημα. Είναι διαφορετικές οι καταστάσεις ανάλογα με τις διάφορες διάφορα τμήματα του στόλου μας και τις διάφορες περιοχές. Και επειδή η μελέτη νομίζω θίγει και κάτι ε, ακόμα. Μας λέει όχι μόνο αυτό που ανέφερα, αλλά ότι κάποια τμήματα του στόλου ε, είναι βιωσιμότερα η ρασιτεχνική με βιωσιμότερα αλληλευτικά εργαλεία, άρα έχουν και κερδοφορία. Αυτό Μα οδηγεί σε μια ερώτηση που την είχαμε θέσει και στην προηγούμενη μεταρρύθμιση τη αλληλευτική Πολιτική το 2012 και το είχαμε συζητήσει τότε. Δεν πρέπει να προβλέψουμε ίδιου κανόνε για όλα τα τμήματα του στόλου μα. Γιατί να ε, έχουμε ευνοϊκή μεταχείριση αυτών που είναι βιωσιμότεροι. Ε, τη μικρή κλίμακα, την ερασιτεχνική, την παράκτη αλεία τίθεται και πάλι το ερώτημα. Πρέπει να έχουμε την ίδια μεταχείριση για όλους, ακόμα και αν τα διάφορα τμήματα του στόλου διαφέρουν μεταξύ τους. Πρέπει όλοι να έχουν την ίδια, ε, τα ίδια ωφέλη όταν είναι διαφορετικό το μέγεθος μικρός και μεγάλος. Δεν είναι για τα αποτελέσματα για όλους μικρούς και μεγάλους. Ευχαριστούμε. Κυρία Ζαμέ, αυτή η μελέτη για το μέλλον της κοινή πολιτικής είναι καλοδεχούμενη. Και σε ό,τι αφορά τον αποκλειστικό ανταγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια είναι τα νέα δικηβεύματα σε διεθνές ε, προσκήνιο και λόγω και της οικολογίας. Πρέπει να δούμε ποια είναι το μέλλον αυτού του κλάδου για την οικονομία μας, αλλά και για την διατροφική κυριαρχία και την οικολογική ισορροπία των πόρων. Στη χώρα μου, τη Γαλλία, τα 7 στα 10 ψάρια που καταναλώνουμε είναι εισαγόμενα. Και όπως είπατε, αν οι συλλογικότητες και εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να διατηρηθούν ε, οι κλάδοι αυτοί. Είμαι από το Μεσόγειο και χαίρομαι που ανταγνωρίζετε ότι έχουμε ξεχάσει ε, την αλία ε, και την καταστροφή στη Μεσόγειο και που πλέον κρούεται τον κόδωνα του κίνδυνου. Αυτό είναι πολύ θετικό. Έχει γνωρίσει τα ωριά της αυτή η πολιτική τη Μεσόγειο, όμως στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου πριν. Η Ιαπωνία είναι στη CGPM. Αλλά ε, λαιλατεί τα χωριτά μας ύδατα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί πρόκειται περί αθέμητου ανταγωνισμού μέσω συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Φυσικά θα πρέπει οι όμορες χώρες να συνεργαστούν με βάση την αρχή της εθνικής κυριαρχίας. Υπάρχουν έλεγχοι, περιορισμοί και πολλοί άλλοι παράγοντες που επιβαρύνουν τους αλληλείς στη Μεσόγειο. Και έχουμε και την ερασιτεχνική αλία, μικρής κλίμακας παράκτια αλία, που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Φυσικά και θέλουμε να υποστηρίξουμε τους μικρούς αλείς, την παράκτια αλία. Τι κάνουμε απέναντι στους ε, μεγάλους όμως ε, παίκτες, ε, τις, τους μεγάλους τόλους ή μεγάλες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται, σέβονται. Δεν πρεονίζουμε το κλάδι πάνω στο οποίο καθόμαστε. Και μην αφήνουμε οικονομίες από την άλλη άκρη του κόσμου να καταστρέφουν τη δική μας. Μου το έλεγε και ένας ψαράς από την περιοχή μου πριν από λίγο καιρό. Ότι τη Μεσόγειο, ε, ε, στη Μεσόγειο παρακολουθούνται πολύ πιο στενά οι ψαράδες από ότι διακινητές είναι άδικο. Δηλαδή κάνουμε επίδειξη ισχύω ε, με τους αδυνάτους και αφήνουμε τους άλλους, τους ισχυρούς. Νομίζω πρέπει να ξαναδώσουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να βάλουν τον κοινό νου εκ νέου στην αλληλευτική πολιτική και στις σχέσεις, και φαντάζομαι συμφωνείτε όλοι, με τις όμορες χώρες τις χώρες ιδίως που έρχονται από τη Μεσόγειο, για να υπάρξει η ισορροπία των ελευτικών πόρων και μια άλλη Μεσόγειος, εν κατακλείδη. Um, Σας ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση. Τη διάβασα αυτή την έκθεση. λέτε για τη Μαύρη Θάλασσα που μαζί με τη Μεσόγειο παραδοσιακά παραγνωρίζονται από την κοινελευτική πολιτική και διέπονταν από δικούς τους κανονισμούς και πολλαπλά στρώματα λήψη αποφάσεων. Και εδώ έχουμε το πρόβλημα με την αηφορία και τον αθέμητο ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, με τα νούμερα που βλέπω, 85% των αποθεμάτων που έχουμε μελετηθεί σε Μαύρη Θάλασσα και Μεσόγειο γίνονται ε, με υπεραλίευση χωρίς ε, βιώσιμο τρόπο δύο-τρεις φορές παραπάνω από τα μέγιστα ποσοστά απόδοσης. Και υπάρχουν και πολλές διμερείς και περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως είπατε για την περιοχή όμως πρέπει να υπάρξει παρόλα αυτά ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ε, θαλάσσια οικονομική ανάπτυξη της Μαύρης Θάλασσας. Γι' αυτό και η διαχείριση της αλίας αυτή την περιοχή μέχρι στιγμής δεν έχει λειτουργήσει επαρκώς. Πότε θα μπορούσαμε να περιμένουμε ένα τέτοιο στρατηγικό πλαίσιο περιεκτικό. Μήπως επίσης έχετε να μας πείτε κάτι για το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη και πιο βιώσιμη διαχείριση της Μαύρης Θάλασσας. Ευχαριστώ για να το ξέρετε, την επόμενη εβδομάδα η Κομισιόν θα μας κάνει μια παρουσίαση ακριβώς γι' αυτό, για τα αποθέματα στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Εσείς κύριε Ντεβίτο. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο κύριος Μπιτό. Σήμερα μιλάμε για τη διαχείριση, την καλύτερη διαχείριση των αλληλευτικών πόρων Μιλάμε για υπεραλίευση. Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση όμως μεταξύ των εφαρμορφών αλίας. Όταν μιλάμε για την κοινή πολιτική αλίας και ευρωπαϊκά κονδύλια και ταμεία, όπως αυτό για την αλία, νομίζω ότι τις προσπάθειές μας θα πρέπει να τις προσανατολίσουμε στους αλίες ε, που ουσιαστικά είναι οι θεματοφύλακες ε, της καλής ε, θαλάσσιας, ε, της καλής κατάστασης των θαλασσών και να τους φροντίσουμε ακριβώς. Μην περιπλέκουμε τους κανόνες και τους βάζουμε παραπάνω εμπόδια και δυσκολίες. Πρέπει να έχουμε όμως μια, μια συνολική προσέγγιση, μιλάμε για υπεραλίευση, μιλάμε για δυσκολίες εξέπρεση αλληλευτικών πόρων. Σε αυτή τη μεγάλη Ευρώπη δεν θα έπρεπε επιτέλους να τα δούμε λίγο πιο σφαιρικά τα πράγματα και να είναι συνεκτικές οι δημόσιες πολιτικές. Έδειξαν και οι τελευταίες ευρωεκλογέ την προσήλωση των Ευρωπαίων στις προκλήσεις του κλίματος, βιοπικιλότητας, της επερθένωση του πλανήτη, συνολικά. ούτε η θάλασσα φεύγει, ε, βγαίνει εκτός της προβληματικής αυτής τα οικοσυστήματα, η θαλασσικό είναι οι πρώτοι που απειλούνται, δυσκολεύονται. Και το ίδιο και συμβαίνει με τα ηχθιαποθέματα. Βλέποντας λοιπόν την ανάγκη να είναι συνεκτικές οι δημόσιες πολιτικές, πρέπει ταυτόχρονα να ξέρουμε ότι ό,τι πάει στη θάλασσα έχει πέρασει από τη γη, από το έδαφος. Υπάρχουν σε επαρκείς ποσότητες ύδατα για να φτάσουν ε, να τροφοδοτήσουν ε, τα μους και τις θάλασσες. Και το νερό που φτάνει και καταλήγει στη θάλασσα είναι καλό ποιοτικά. Σήμερα οι δημόσιες πολιτικές της Ένωσης δυστυχώς ευνοούν ένα εντατικό γεωργικό μοντέλο με χρήση ε, που φτάνουν και όλα αυτές οι τοξικές ουσίες φτάνουν στη θάλασσα. και αποδυναμώνουν ε, τους ε, λευτικούς σπόρους. Ας μην δείχνουμε λοιπόν και καταλογίζουμε τα πάντα στους αλείς. Ας πιάσουμε το θέμα πιο νωρίς στην πηγή του. να φροντίσουμε το περιβάλλον και την κατάστασή του για να μπορέσει να αποκατασταθεί και ο αλληλευτικός πλούτος. Μιλήσατε επίσης για την οικονομική ευρωστία κάποιων επιχειρήσεων, που είναι όλο και μεγαλύτερη. Ναι. Έχουμε και το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Ε, όταν είναι λίγη προσφορά αυξάνονται οι τιμές. Ε, και ισχύει αυτό με κάποια λιεύματα. Εγώ όμως θεωρώ ότι ε, υπάρχει ο κίνδυνος η αλία να πεθάνει υγιέστατη παρόλα αυτά. Δηλαδή, να πετύχει εγχείρηση αν πεθάνει ασθενή. Άμα χαθούν οι πόροι και αν δεν τα φροντίζουμε τα πράγματα ανάντι, κάποια στιγμή θα αφανιστεί αυτή η δραστηριότητα. Και όσοι ζουν ακόμα θα το δουν. Μια υγιέστατη δραστηριότητα παρόλα αυτά να πεθαίνει. Well, thank you very much. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Καθηγητά Λεγκαλίκ. Ε, Ακούσαμε διάφορες ερωτήσεις, δεν υποχρεούστε βεβαίως να απαντήσετε απολύτως τα πάντα, αλλά εγώ έχω μια πρόσθετη ερώτηση. Γιατί στο Λουξεμβούργο τρώτε τόσα πολλά ψάρια? Bien. <clears throat> Merci, euh, Monsieur le Président. Euh, je malheureusement Πρόεδρε, δυστυχώ δεν έχω στοιχεία στη διάθεσή μου για να μπορέσω να απαντήσω στην τελευταία σας ερώτηση. J'imagine Εμείς έχουμε στοιχεία συνολικά για τα νοικοκυριά και σχετικά με τα νοικοκυριά του Λουξεμβούργου είναι περιορισμένες οι πληροφορίες μας. Τώρα, κάποια γενικά στοιχεία. Να ξεκινήσω από το τελευταίο που ανέφερε ο κύριος Μπιτού. Ίσως να το ακούσουμε και στην επόμενη παρουσίαση, αλλά δεν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση σήμερα κατά την οποία έχουμε μια επιδίνωση των Αντίθετα έχουμε μια συνολική βελτίωση. Προφανώς έχουμε κάποιες περιοχές κρίσιμες όπου χρειάζονται βελτιώσει, αλλά σε σχέση με πριν από 15-20 χρόνια υπάρχει μια συνολική βελτίωση, συνολική και γενική, της κατάστασης του αποθέματος. Για τα κοχύλια, ε, τα κοχύλια Σανζάκ τέλος πάντων, αυτά αλλιεύονται κατά τρόπον ώστε να διατηρείται περίπου ο αριθμός των σκαφών που προβαίνει σε αυτήν την ειδικευμένη δραστηριότητα και με συγκεκριμένη αδειοδότηση. Και μιλώ για βελτίωση και των οικονομικών επιδόσεων στην λεγόμενη βιομηχανική κλίμακα αλληλεία έχουμε ήδη τοπικά ε, που έχουν υψηλότατο δίκτυο κερδοφορίας. Υπάρχει λοιπόν μικρότερος όγκος αλλιεύματος, αλλά σε υψηλότερη και πιο κερδοφόρα τιμή. Concernant la Για την πρώτη ερώτηση που έθεσε η κυρία Αγγιλέρα με σχετικά με τον αντίκτυπο της οδηγίας επί των συνδικών εργασίας είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην περαιτέρω αύξηση του διαφορικού ανταγωνιστικότητος μεταξύ των Ευρωπαίων αλλιέων και των μη Ευρωπαίων αλλιέων. Ιδιαίτερα για διεθνοποιημένες, παγκοσμιοποιημένες αγοράς, όπως, αγορές όπως αυτές των θηνοειδών, του τόνου. Με τελείως διαφορετικές συνδίκες εργασίας και τελείως διαφορετικό εξοπλισμό και προϋποθέσεις. Αυτό μπορεί να έχει σημαντικότατο αντίκτυπο επί της ανταγωνιστικότητας του ενωσιακού τομέα. Για τις προστατευμένες προελεύσεις και την αναφορά τους ως ε, έναν τρόπο προαγωγής, προώθησης των ε, αλλιευτικών προϊόντων. Σε πρόσφατη μελέτη είχαν καταλογοποιηθεί 50 συνολικά περίπου είδη για τα οποία μπορούσε, υπήρχε ένας τρόπος τέτοιας επισήμανσης, το οποίο βεβαίω χρειάζεται και ένα χρόνο για να αναπτυχθεί, αλλά πράγματι επιτρέπει στον καταναλωτή να έχει πρόσθετη και πλήρη πληροφορία και ενημέρωση. για τις δυνατότητες ίσως δημιουργίας ενός σήματος για το σύνολο των προϊόντων, αυτό συνήθως μπορεί να γίνει για τα νοπά προϊόντα, αλλά δημιουργεί σημαντικά προβλήματα για τα μεταποιημένα. Διότι υπό τους κανόνες του, του διεθνούς εμπορίου θα έχουμε προϊόντα που μπορεί να είναι made in France ή made in Germany τέλος πάντων αλλά που μπορεί να περιέχουν και στοιχεία από άλλες χώρες και από παντού στον κόσμο. Και επομένως θα είναι δύσκολο να έχουμε μια πλήρη ενημέρωση για την προέλευση του αρχικού προϊόντος, λέει ο μιλητής. Αλλά θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάτι τέτοιο, όπως το είχαμε κάνει και πριν από χρόνια εξετάζοντας ακριβώς την έννοια, το σκεπτικό του τι σημαίνει made in τάδε χώρα. Αυτό που αναφέρθηκε επίσης για τις, ε, τα θεσμικά εστιατόρια, καντίνες και τα λοιπά, ε, στην καλήθεια ε, είχε γίνει αυτό τα πλαίσια της προώθησης ε, κάποιων τοπικών προϊόντων και κάποιων δήμων στη Γαλλία που θα πρότειναν στις σχολικές τους ε, ε, καντίνες να έχουν αντίστοιχα τοπικά προϊόντα τοπικής προέλευσης αυτά τεχνικώς είναι πραγματοποιήσιμα, υλοποιήσιμα. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο σήμερα για έναν διαχειριστή εστιατορίου να παραγγείλει ένα ψάρι ε, από τον Ειρηνικό τρεις μήνες νωρίτερα παρά να βασανίζεται για να βρει τα τοπικά προϊόντα. Βεβαίω δεν, θα δεν θα υπήρχε το κόστος κατάψυξης και μεταφοράς ενδεχομένως έχει κάποιες δυσκολίες και προϋποθέσεις και απαιτήσει, αλλά τεχνικός μπορεί να γίνει. This is a good time for me, uh, Professor ε, καθηγητά Λογκαλίκ, ε, ε, νομίζω ότι έχουμε, εγώ δηλαδή, εγώ φταίω, ε, ξεχάσαμε λίγο το χρόνο και πρέπει να συντομεύσουμε. Μάλιστα, Πρόεδρε, για τον κύριο Φερέιρα, και ίσως αυτό σχετιζόταν και με άλλη ερώτηση, για τις ελεύθερες συναλλαγές είναι πολύ σημαντικό να δει κανεί ποιες είναι οι πρακτικές των προϊόντων των αλλιευτικών και της υδατοκαλλιέργειας με τις χώρες εκείνες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επιθυμεί να συνάψει τέτοιες σχέσεις συναλλαγών. Γιατί αυτό θα μπορούσε να έχει ταχύτατα πολύ αρνητικές συνέπειες επί της ανταγωνιστικότητας του τομέα του συγκεκριμένου. Μπορούμε να αναλαμβάνουμε μέτρα εμπορικά όταν έχουμε ταυτοποιήσει, εντοπίσει συγκεκριμένες πρακτικές ή προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί υπό συνθήκες που δεν, είναι, δεν συμμορφούνται προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, με αυτό ολοκληρώνω. Σας ευχαριστώ και εγώ λέω Πρόεδρε. Πάμε στο επόμενο σημείο της παρουσίασης. Η κυρία Ούλριχ. Regardez ma présentation, s'il vous plaît. Donc, je vais parler aussi en... Θα μιλήσω και εγώ γαλλικά. Περιμένω βέβαια να ξεκινήσει. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αγαπητοί βουλευτέ. Επανέρχομαι στο ένα για τη διαχείριση αλίας δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα ένα που με απασχολεί. Για να δω. Μπορώ να αλλάζω διαφάνειες από εδώ. Λοιπόν, διάλεξα να ξεκινήσω με κάποιες ε, εικόνες που τις έχω ξαναδείξει στο προηγούμενο κοινοβούλιο για να θυμίσω ποιες είναι οι βασικές αρχές ε, της ε, διαχείρισης σε ό,τι αφορά την μέγιστη βιώσιμη απόδοση, γιατί εκεί βασίζονται και όλες νομίζω οι ερωτήσεις που ετέθησαν και βοηθάει να καταλάβουμε το βιολογικό οικολογικό πλαίσιο, διότι όλα τα θέματα και δυσκολίε από εκεί απορρέουν, από την οικολογική πολυμορφία και διαφορετικότητα στην αλία σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, ε, η βιολογία είναι πολύ απλή, ότι αν δεν υπάρχουν ε, πολλά ψάρια δεν αναπαράγονται πολύ και δεν κερδίζουμε και πολλά σε ό,τι αφορά την αλία. Όσο περισσότερο αυξάνεται ο όγκος των ψαριών στη θάλασσα, τόσο περισσότερο παράγονται πρωτεΐνες και νέα ε, ψάρια γεννιούνται καθημερινά, πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός λοιπόν, αυξάνεται και έχει τη μεγαλύτερη αύξηση και παραγωγικότητα. Ενώ ε, όταν φτάσει το φυλαλίδιο αυτό να γεμίσει, σταματάει η ανάπτυξη και μένουμε σε χαμηλά επίπεδα απόδοση, γιατί υπάρχει περιορισμένο χώρο ή περιορισμένη τροφή. Άρα, ποιο είναι ο στόχο τελικά τη βιώσιμη ανάπτυξη, ε, να έχουμε ε, τη δυνατότητα να στο πλέον παραγωγικό τη επίπεδο την. Ε, μάλλον διότι διατηρηθεί στο το επίπεδο των πληθυσμών των ψαριών. Αυτό είναι ο στόχο τη μέχρι βιώσιμη απόδοση, μια σταθερή ισορροπία μεταξύ παραγωγικότητα ενό πληθυσμού, το μέγεθο του γλυκού, αν θέλετε, και του αριθμού των αλλιών, αυτών δηλαδή που θα μοιραστούν το γλυκό, την πίτα. Και πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ φύσης και εκμετάλλευσης. Στην πραγματική ζωή όμως που δεν είναι φιαλίδιο, δεν είναι μια γυάλα με χρυσόψαρα ή άλλα ψάρια, ε, δύσκολα μπορούμε να βρούμε αυτή την ισορροπία που μπορούμε να πετύχουμε μέσα σε αυτή τη γυάλα. Αλλάζει θερμοκρασίες, οι άλλες καιρικές συνθήκες, το πλακτόν, ε, τα αριθμό των ψαριών, ε, έχουμε αρπακτικά επίσης, ήδη και όχι μόνο τους αλείς που πάνε να φάνε τα ψάρια και έχουμε και τι διάφορες μορφές αλήθεια, τα διάφορα ληφτικά εργαλεία κτλ. Άρα το θαλάσσιο περιβάλλον συνεχώς αλλάζει. Είναι ένα είδο ιερού γκράλ, ένα είδο του. Δύσκολα μπορούμε να το εντοπίσουμε, ε, να το βρούμε. Και πολλές φορές ε, το βλέπουμε αφού το χάσαμε. Ε, αλλάζουν τα πράγματα λοιπόν, τα πάντα ρί. Και είναι δύσκολο να τα προβλέψουμε. Αυτή λοιπόν η διαφορετικότητα κάνει και τόσο δύσκολα διαχειρίσιμη την αλληλεία. Αυτά νομίζω τα βασικά έπρεπε να σας τα υπενθυμίσω. Ο Μπερτρόν σας έκανε μία παρουσίαση. Υπήρξε πρόοδος Πάντα έχουμε μια πολύ αρνητική εικόνα για την αλία, ότι τα ε, πράγματα πάνε πολύ άσχημα, δεν έχει μείνει ψάρι ούτε για δείγμα. Όχι όμω. εδώ για 15 χρόνια στην Ευρώπη υπήρξε πρόοδο. Βλέπω λοιπόν σε αυτό το γράφημα ποια είναι η πρόοδος των αποθεμάτων. Ποια θεωρούνται ότι ε, είναι θύμα υπεραλίευσης. Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς μας το 5%. Δηλαδή μπορούμε να το δούμε μισό άδειο, μισό γεμάτο το ποτήρι και σε ό,τι στη βιώσιμη απόδοση. Άλλοι θεωρούμε ότι πλησιάζουμε, άλλοι θεωρούμε ότι δεν πλησιάζουμε. Ε, πάντως είμαστε και στο 5%. Προς τα κάτω βλέπετε τη βιομάζα. Ε, τα ψάρια αυτά δεν τα συζητάμε και πολύ. Οι δύο καμπύλες από πάνω, ιδίω ε, ατλαντικός και εξωτερικές ε, ζώνες πλην ένωσης, δηλαδή παραδείγματος χάρη με Νορβηγία ή νησιά Φερόε, εκεί έχουμε αύξηση. Άρα κατά μέσο όρο τα αποθέματα, τα ευρωπαϊκά, στον Ατλαντικό έχουν αυξηθεί κατά 40% σε βιομάζα εδώ και τα τελευταία 15 χρόνια. Στο βάθος, μάλλον οι χαμηλές καμπύλες είναι Μεσόγειος ε, και η Μαύρη Θάλασσα. Δεν έχουμε μεγάλη βελτίωση εδώ. κάπου αρχίζει όμως ε, ε, γιατί γίνονται πολλά πράγματα στη Μεσόγειο, θα επανέλθω όμως. Κρατήστε αυτή την εικόνα. Δεν είναι τόσο μαύρο-άσπρο. Είναι λιγότερο αρνητικά τα πράγματα σε σχέση ίσως με την εντύπωση που κανείς ε, αποκομίζει αν διαβάζει τον τύπο ή ε, βλέπει τηλεόραση. Ποιοι είναι οι στόχοι του 13. Και μια μείζων πρόκληση που δεν την έχουμε πετύχει είναι υποχρέωση εκφορτώσεων, μιας απορρίψεων. Η Ευρωπαϊκή Αλιά παράγει, μάλλον ε, κάνει πολλές απορρίψεις και μετά το 2015 δεν είχαμε μεγάλη πρόοδο. Το πρώτο σχήμα εδώ που βλέπετε είναι οι αναφορές που στέλνουν κάθε χρόνο τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς έχουν βελτιώσει την κατάσταση με τις εκφορτώσεις το ΣΤΕΣΦ ε, τα παρακολουθεί και δείχνει την κατάσταση σε κάθε χώρα. Περισσότερη εφαρμογή, μεγαλύτερη βελτίωση δηλώνουν τα κράτη-μέλη ή όχι σε ό,τι αφορά τις εκφορτώσεις. Βλέπετε ότι ε, λίγα πράγματα έχουν γίνει. Στην αρχή κάτι έγινε, αλλά η οχι σε οτι αφορα εκφορτωσεις βλεπετε είναι πενιχρή. Και κάποιες χώρες μόλις αρχίζουν να υλοποιούν τα υπεσχημένα υπήρξε μεγάλη αντίσταση από τους ψαράδες και τη βιομηχανία σε αυτό τον κανονισμό. Σε ό,τι διάφορα πληροφόρηση και ενημέρωση για τα λιεύματα, εδώ έχουμε και οπισθοδρόμηση. Για μας τους επιστήμονες που χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ψαριών που αλλιεύονται, έχουμε οπισθοχώρηση. Βλέπετε εδώ σε αυτό το σχήμα που βρισκόμαστε, ποιες είναι οι τελευταίες προφορίες. Ε, με το γαλάζιο έχω επιλέξει τη Βαλτική. Βλέπετε τις απορρίψεις ε, που εκφορτώνονται και πολλούνται. Και με το κόκκινο βλέπετε τις εκτιμήσεις ε, των βιολόγων για τους πραγματικές απορρίψεις. Δηλαδή βλέπετε πόσο πιο ψηλά είναι τα κόκκινα, οι πορτοκαλί, οι πορτοκαλί από τις μπλε. Ενώ εμείς θα θέλαμε να εξαφανιστεί το κόκκινο και να βλέπουμε μόνο μπλε. Έχω τώρα διαλέξει τρεις μελέτες περιπτώσεων. Είναι ίσως πιο προβληματικές περιπτώσεις, όχι απελπισμένες, αλλά τέλος πάντων απελπιστικές μάλλον, αλλά εκεί που η επίτευξη των στόχων υστερεί περισσότερο και είμαστε απεσιόδοξοι για το κατά πόσο θα το καταφέρουμε στο μέλλον. Πρώτη περίπτωση είναι ο γάδος στη Βαλτική που ακούστηκε πολύ. Αν δείτε την εθνιτότητα και τη βιομάζα, βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη διακύμαση στο αποθέματο στα τελευταία 20 χρόνια, έχει σκαμπανεβάσματα. Αλλά από κοντά αν το δούμε, ο πληθυσμό αυτό οικολογικά υποφέρει και βιολογικά. Η μπορεί να είναι μεγάλη ε, σε μέγεθος. Εδώ βλέπω ότι είναι όλο και πιο μικρή και αδύνατη. Βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία. Σαν σαρδέλα μοιάζει αυτός ο μπακαλιάρος. Επίσης ε, είναι ένα ψάρι πολύ ευάλωτο ε, σε πτές από παράστα. Εδώ βλέπετε το ε, το, το σηκώτη ε, του βακαλάου. Ε, οι φώκες επηρεάζουν πολύ την κατάσταση εδώ. Και τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ ώστε να νιώθουμε σχεδόν απελπισμένοι ότι θα καταλήξουμε στα επίπεδα του παρελθόντος. Μπορεί πριν από 10, 15, 20 χρόνια να είχαμε αλλιεύσει λιγότερου μπακαλιάρου. Θα είχαμε καλύτερη κατάσταση τώρα. Δεν ξέρουμε. Δεύτερο παράδειγμα, στην Αδριατική, ο γάβρο και η σαρδέλα, που είναι τα βασικά αλλιεύματα τη Μεσογείου. Εδώ ε, υπάρχει μια δυσκολία να εκτιμήσουμε από επιστημονικής και βιολογικής πλευράς το αν τα αποθέματα αυτών των ψαριών αυξάνονται ή μειώνουν ποια είναι η μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Δεν καταλήγουμε σε επιστημονική συνένεση. Αυτά είναι τα τελευταία αποτελέσματα για την κατάσταση των αποθεμάτων. Από το 17 και μετά δεν έχουμε στοιχεία. Και στο πρώτο γράφημα, πάνω αριστερά, είναι η αύξηση της συντότητας ανά είδος και η εξέλιξη των αλληλευμάτων τα τελευταία χρόνια. Μεγάλη μείωση. Βλέπετε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, χωρίς να ξέρουμε όμως ακριβώς ποια είναι η κατάσταση. Πρέπει να υπάρξουν πραγματικές πολιτικές ε, διαχείρισης για τα αποθέματα αυτά που δεν είναι αντικείμενο καλής διαχείρισης. Τρίτη περίπτωση, βορειοδυτικά νερά, κελτικό πέλαγος, ιρλανδικό πέλαγος, ε, εκεί γύρω από τη Σκοτία μικτή, μεικτά αλλιεύματα. Κάποια πάνε καλά, κάποια δεν πάνε. Και εδώ έχουμε μεγάλη δυσκολία να βρούμε μια ισορροπία με όλα αυτά τα αποθέματα. Και χρησιμοποιείται πολύ ο όρος choke species, δηλαδή τα είδη παγόμενα σε περιοριστική ποσόστοση. Δηλαδή ή είναι πολύ χαμηλή η ποσόστοση και άρα υπάρχει υπεραλήψη ή υπάρχει πολύ κακή κατανομή των ποσοστώσεων. Δηλαδή κάποιες χώρες έχουν μεγάλες ποσοστώσεις, μεγάλο μερίδιο της ποσόστοσης και άλλες τίποτα. Και έχουμε πολλές απορρίψεις. Αυτή είναι η μελέτη που έγινε πριν από 2-3 χρόνια για τα διάφορα αποθέματα που κινδυνεύουν περισσότερο. Βλέπετε, έχουμε μία σύγκρουση ε, για το τι πρέπει να αλλιεύεται και το τι αλλιεύεται. Αυτά για το Ιρλανδικό ε, πέλαγος και για τη Δυτική Σκοτία. Πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, ιδίως τώρα, γιατί για κάποια ε, υπάρχει η σύσταση να μην αλλιεύονται καθόλου κάποια αλλιεύματα. Αυτό όμως δεν γίνεται. Άρα υπάρχουν ασυγκρόμενοι μεταξύ τους και αντιπαρατηθέμενοι μεταξύ τους στόχοι. Ποιες είναι οι προκλήσεις ε, για την αλληλεία. Πρώτον, τι μπορούμε πρώτα να κάνουμε σε ό,τι αφορά την υποχρέωση εκφορτώσεων και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Αν δείτε κανεί τι αναλύσει έγιναν, στο βορειοδυτικό έχουμε τώρα 15 τη κοινή αλληλευτική πολιτική που προτείνει κάποιε προσαρμογέ. Δεν χρησιμοποιούνται κάποια μέτρα από αυτά που έχουν προταθεί, οι άλλα χρησιμοποιούνται μένα, αλλά δεν είναι αποτελεσματικά δε. Άρα δεν βοήθησε την υλοποίηση και τη βελτίωση κατάσταση ε, η νομοθεσία Ποιο είναι το μείζον θέμα για το οποίο μιλάμε συνεχώ, όπω στον κώδικα οδική κυκλοφορία, χρειάζεται περισσότερο έλεγχο. Τι λέει ο κώδικα οδική κυκλοφορία. Ανεξαρτήτω το αν ένα αυτοκίνητο είναι μεγάλο ή μικρό, δεν πρέπει να κάνει υπέρβαση του όριου ταχύτητα και βάζουμε κάμερε για να τη, ε, το όριο ταχύτητα. Είναι επίμαχο ε, το θέμα, αλλά όταν εφαρμόστηκε το όριο ταχύτητα και το ραντάρ απέριξε. Βλέπετε εδώ. Δεν κοιτάμε τον Αλιέα, τον Ψαρά, αλλά τι περνάει. Και βλέπω, τεχνολογική πρόοδος ε, βοήθησε στην αυτοματοποίηση και στην πολύ γρήγορο εντοπισμό των ειδών τα οποία αλλιεύονται. Δανία. Έχω εργαστεί εκεί 20 χρόνια. Είναι σε πολύ προηγμένη φάση. Βλέπετε εδώ έναν ε, ψαρά που συμμετείχε στις έρευνες αυτές. Εδώ βλέπετε για κάθε μέρα αλίευσης. Τι αλίευε, μικρά, μεγάλα ψάρια. Τα μικρά είναι τα κίτρινα, Ούτε ένα δεν βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία. Από τη μια μέρα στην άλλη που έχει κάνει προσπάθεια με την κάμερα ο Ψαράς, ε, την, ε, από τη μια μέρα στην άλλη όμως άρχισε να εκφορτώνει και όχι να απορρίπτει τα μικρά ψάρια. Άρα περισσότερος έλεγχος, περισσότερα κίνητρα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αλία. Βελτιστοποιείται η ποσόστοση πολύ θετικά τα, τα παραδείγματα από, αυτή την, από αυτό το μέτρο. Δεύτερη πρόληψη. Έπρεπε να προσθέσω εδώ τη Μεσόγειο, συγγνώμη, την ε, Μαύρη Θάλασσα. Ε, έχουμε τη Μεσόγειο, Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα. Πολύ μικρά σκάφη. Επίσης, το πρόβλημα είναι η πίτα. Δεν είναι παραγωγική Μεσόγειος, είναι αρκετά φτωχή ε, πολύ λίγο οξυγονώνεται, είναι πολύ αλμυρή ε, και άρα τα ψάρια δεν είναι και τόσο παραγωγικά. Υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα εδώ ανάμεσα στον αριθμό των αλιέων και τον αριθμό των ψαριών. Δύσκολα μπορεί κανείς να βρει μια ισορροπία μεταξύ του κοινωνικο-οικονομικού αντικτύπου και της οικολογικής παραγωγικότητας της Μεσογείου που είναι πολύ μικρή. Και όπως ξανάπα πριν, για πολλά χρόνια η Μεσόγειος ε, είχε εγκαταλειφθεί, η διαχείριση ήταν ελάχιστη. Εδώ και τρία χρόνια περίπου έχουν αλλάξει τα πράγματα και γίνεται μια πραγματική προσπάθεια από τις μεσογειακές χώρες. Medfish Forever είναι αυτή η δυναμική που εφαρμόζεται και στην ε, Μαύρη Θάλασσα επίσης για να αλλάξει η κατάσταση. Οι προτεραιότητες λοιπόν εδώ από τις μεσογειακές χώρες τα από Μπερτρά εν ολίγης, είναι η καταπολέμηση της ε, παράνομης αλίας, που είναι ένα μείζον ε, στοιχείο που μπορεί να βελτιώσει και να οδηγεί σε προστασία των θεποθεμάτων. Ε, και το δεύτερο είναι η προστασία με βιώσιμο τρόπο της αλίας μικρής κλίμακας. Κάνει πολλά η ΦΑΟ στην Μεσόγειο και αλλού για να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ ψαράδων και ψαριών στην αλία μικρής κλίμακας. Επόμενη, έχουμε αύριο την έκθεση στο IPCC. Κλιματική αλλαγή πραγματικά διαταράσει και φέρνει τα πάνω κάτω σε όλα όσα σας είπα. Η ΦΑΟ κάνει πολλά και εδώ για να προκαταλάβει την επίπτωση που θα έχει η κλιματική αλλαγή στις στοχότερες ε, περιοχές του κόσμου. Εμεί στην Ευρώπη που είμαστε στη μέση ουσιαστικά. Δεν θα χάσουμε τα περισσότερα εμείς. Ε, βλέπετε ότι στη... αυτές που απληγούν θα είναι οι τροπικές, οι κόκκινες αυτές εκεί στο χάρτη χώρες. Ε, όχι οι βόρειε. Ε, Νορβηγία, Ισλανδία. Ε, ωφελούνται κιόλας από την κλιματική αλλαγή. Αλλά ένα σημαντικό είναι να πούμε ότι χάνουμε σε παραγωγικότητα με την κλιματική αλλαγή, αλλά στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να κερδίσουμε κάποια παραγωγικότητα αν διαχειριζόμασταν τώρα τη μέγιστη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό προσπα... Απόδοση. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Ότι ναι, μεν η παραγωγικότητα μειώνεται, αλλά αν έχουμε καλή διαχείριση θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του γραφήματος σε μπλε και σε κόκκινο. Τι ήθελα να σας πω συμπεράσματα. Η διαχείριση αλλίας πράγματι είναι κάτι δύσκολο, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ε, τα ψάρια μετακινούνται, δεν τα βλέπουμε και δεν μπορούμε να προβλέψουμε πολλά ε, από τα μελλοντικά στοιχεία. Άρα πρέπει αυτή την πολυπλοκότητα να αντιλάβουμε υπόψη και να αντιλαμβάνουμε πάντοτε υπόψη. Τίποτα δεν είναι απλό στην αλληλία. Αν ήταν θα το είχαμε ήδη βρει. Δεύτερο συμπέρασμα, η κοινή ελευτική πολιτική του 13 ήταν ε, μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που γινόταν η διαχείριση. Είχαμε τους στόχους τώρα για την εκφόρτωση, ε, τη μέγιστη βιώσιμη απόδοξη, πολύ καινοτόμα στοιχεία, όμως ακόμα έχουμε να ξεπεράσουμε ιστορικούς θεσμικούς πύχης. Γι' αυτό είναι δύσκολο. Και υπάρχουν και νέες απειλές τον εθνικισμό, για να μην πω Brexit, αλλά τέλο πάντων έχουμε την σύγκρουση με Ισλανδία, Νορβηγία ή τα νησιά Φερόε. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα πρόβλημα και επιχορηγήσει που επανέρχονται στο πολιετέ και στο Τάμι για την Αλία. Το βλέπουμε παντού. Είναι τεκμηριωμένο. Οι επιδοτήσει ε, οδηγούν σε μεγαλύτερη υπεραλίευση και πλεονάζουσα παραγωγή. Άρα, να προσπαθήσουμε να πετύχουμε το, τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση είναι ο βασικός στόχος γιατί ωφελεί τους πάντες, ψάρια, ψαράδες και ασφάλεια επιστηστική. Και ακριβώς λόγω της διακύμασης και της, της ποικιλότητα θα πρέπει να έχουμε μία μακροπρόθεσμη άποψη αλλά να έχουμε υπόψη μας και τι γίνεται με το οικοσύστημα, γιατί είμαστε σε ένα πλοίο μέσα στην τερκυμία αυτή τη στιγμή. Το επόμενο είναι ότι η αλία πρέπει Μάλλον, πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα λεύματα και όχι μόνο όσα εκφορτώνονται. Χρειαζόμαστε καταγραφή όλων και της αεραστεχνικής, ε, μάλλον και των παρεπιπτόντων ε, αλλιευμάτων και όλα να τα περιλαμβάνει. Και να χρησιμοποιούν περισσότερο τα κίντρα που δίνουμε. Υπάρχουν σχάρια για να μπορεί κάποιο να έχει μια εξαίρεση ή μια καλύτερη ποσόστοση. Θα πρέπει να χειρίζεται καλύτερα τα, τις, τα λιεύματά του. Στο άρθρο 15, υποχρέωση εκφορτώσεων, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά με πιο έτσι, θετικό για εμάς τρόπο. Και το τελευταίο στοιχείο, στο πλαίσιο των ε, συστάσεών μου, να προσέξουμε την ε, το πλεονάζον αυτό δυναμικό, να προσέξουμε τις επιδοτήσεις, να προσέξουμε την παράνομη αλία. Και η τελευταία μου λέξη είναι, τα ψάρια είναι παραγωγικά. Αυτό είναι το θετικό. Ποτέ δεν είναι αργά. Και με τα μέτρα μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Κάλλια αργά παρά ποτέ. Και μας το λέει και η κλιματική αλλαγή. Ένα απόθεμα που πλήττεται από υπεραλίευση δεν είναι ανθεκτικό, είναι πολύ ευάλωτο και στο μέλλον θα τα πάει χειρότερα. Άρα, κάλιο αργά παρά ποτέ. Nothing... Ευχαριστούμε κύριε καθηγητρία. Τίποτε δεν είναι εύκολο. Άρα αν ήταν εύκολο δεν το κάναμε καν. Ερωτήσεις. Ναι, ε, μόνο ερωτήσεις. Για την παρουσίασή σας έχω να ρωτήσω το εξής. Για το θέμα των εκφορτώσεων. Είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε το ερώτημα γιατί έχουμε φτάσει εδώ. Δεν έχει εξηγηθεί. Ένα από τα πιο σημαντικά αίτια φαίνεται να είναι ότι η οι αλείς αναγκάζονται να εκφορτώσουν είδη που έχουν αλλιευθεί ως παρεπίμπτοντα αλλιεύματα. Το ερώτημα είναι ποιο από το ποσοστό αυτό επιβιώνει. Και το ερώτημα το δυσκολεύουμε ακριβώ γιατί υπάρχουν υποχρεωτικέ εκφορτώσει. Οπότε έτσι δεν γνωρίζουμε πραγματικά την κατάσταση των αποθυμάτων. Πρέπει όμω να ψάξουμε και λύσει. Τι γίνεται με την ε, αλία εκτό ποσόστοσης. Τι λύση θα μπορούσε να είναι αυτή για τις υποχρεωτικές εκφορτώσεις. Κατά την άποψή σας λοιπόν, η λύση αυτή, η λύση των υποχρεωτικών εκφορτώσεων με παρεκκλήσεις θα ήταν ε, μια οδός που μπορούμε να ακολουθήσουμε Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την καθηγητρία Ούλρικ. Σημειώνω ότι δώσατε ιδιαίτερο βάρος στην παρουσίασή σας στις κλιματικές αλλαγές και στη μελέτη αυτή βλέπουμε ότι ένα μέρος της επιστημονικής κοινότητας θεωρεί ακριβώς ότι η παρθέρμανση του πλανήτη επηρεάζουν πολύ σοβαρά την θαλάσσια ζωή. Ιδίω οι χώρε του Νότου πλήττονται ιδιαίτερω. Και αυτό είναι ένας πολλωστός ε, συναγερμός, ένα κουδουνάκι προειδοποίησης που ακούμε εδώ και καιρό. Δεν είναι απλώς μια πιθανότητα, είναι βεβαιότητα ότι υπάρχει πρόβλημα και για τις θάλασσες. Εάν δεν μπορούμε να προστατεύσουμε την κλωδία και την πανίδα της θάλασσας, ε, πρέπει τουλάχιστον να αναλάβουμε ευθύνες απέναντι στους αλείς μας. Και η ερώτησή μου είναι, προ την ε, καθηγητρία. Υπάρχουν πρόσφατε μελέτε για τον πραγματικό αντίκτυπο στα αποθέματα και το τι γίνεται με τι πετρελοκυλίδε. Με την ρήπανση από τα ζωτούχα και τα μικροπλαστικά επίση. Ε, αναφέρατε ότι οι επιδοτήσει ε, έχουν οδηγήσει σε υπερπαραγωγή. Μπορείτε να το εξηγήσετε καλύτερα, διότι αν θυμηθώ, αν σκεφτώ μάλλον, τι γίνεται με τις χρηματοδοτήσεις για τους δικούς μας τους αλείς, που έχουν να αντιμετωπίσουν περιόδους ε, πάυσης της αλληλευτικής δραστηριότητας ή μέτρα για τον εξοπλισμό των σκαφών τους ώστε να γίνουν ασφαλέστερα. Δεν το κατανοώ ακριβώς όπως εσείς. Εσείς μπορείτε να μου το εξηγήσετε καλύτερα και το δικαιολογήσετε. Πώς ακριβώς έχει ευνοηθεί η υπερπαραγωγή. Ο κύριος ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι οι, οι πληροφορίες αυτές που λαμβάνουμε μπορούν να μας βοηθήσουν να χαράξουμε καλύτερα την μεταρρύθμιση των πολιτικών που μας απασχολούν και ήταν διαφωτιστική η παρουσίαση που ακούσαμε εδώ, καθώς είναι και μελέτη η ερμηνεία βέβαια μετά από μια ανάγνωση της μελέτης μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από τον καθένα και να προκύψουν και αντιφάσεις. Είναι προφανές ότι πρέπει να ελέγξουμε την αλία, ιδίω στο πλαίσιο της αβεβαιότητας, της αβεβαιότητας που επικρατεί για το μέλλον των ωκεανών. Ε, είναι τεράστια κλίμακα όσων συμβαίνουν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι κλιματικές αλλαγές έχουν πολλαπλές πτυχές που θα επηρεάζουν όλο και περισσότερο τη θαλάσσια ζωή, ιδίω τα είδη που μα ενδιαφέρουν. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα ήθελα να είμαι αισιόδοξο. Για την Αλία, ε, νομίζω ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την Αλία στην Ευρώπη και την επιβίωση των ειδών μέσω κάποιων στοιχείων που είναι και θετικά. Για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα βεβαίως αυτό είναι ουσιώδες αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι μπορούν ε, να επιβιώσουν και οι κοινότητες αλλιέων, δηλαδή βιωσιμότητα και για αυτές τις κοινότητες. Σήμερα ο μέσος όρος ηλικίας των Ευρωπαίων αλλιέων είναι περίπου 50 ετών. Όλο ένα και λιγότεροι προσελκύονται από την αλλία, οι νέοι δηλαδή. Είναι και δύσκολη η αλία και επικίνδυνη. Οπότε η ερώτησή μου είναι, ακούσαμε πολλά για τις εξελίξεις. Είναι αναπόφευκτο. Επιδοτήσεις για τον εξυγχρονισμό του στόλου οδηγούν αναπόφευκτα σε υπεραλίευση. Μήπως εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο συγκρατημένη ε, προσέγγιση, γιατί είναι πιο διαφοροποιημένη η πραγματικότητα. Σε κάποιες κοινότητες αλλιέων με ερασιτεχνικότερη δραστηριότητα είναι καθοριστική σημασία η ενίσχυσή τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν, να παραμείνουν βιώσιμες δηλαδή και να παραμείνουν ασφαλή και τα σκάφη τους. Χρειάζονται όμως και νέες γενιές ψαράδων για μια δραστηριότητα που είναι ουσιώδου σημασία για την Ευρώπη και για την επιβίωση συγκεκριμένων κοινοτήτων. Την ερώτηση αυτή την αντιστρέφω προς την ε, υποψήφια πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είπε ότι ναι, πρέπει να εκπαιδεύσουμε νέους ψαράδες ε, στην Αλία και να βάλουμε και τουαλέτες στα σκάφη και Wi-Fi. Αστείο ήτανε. Κύριε Φερέιρα, σας προειδοποιώ, θα σας προσπαθήσω να σας περιορίσω στα δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ένα από τα θέματα που σχετίζεται και με το τελευταίο. Δεν κατανοώ τον συσχετισμό, τον αυτόματο συσχετισμό χρηματοδότηση-επιδότηση και υπεραλίευση. Δεν πρέπει να γίνεται αυτή η εξίσωση. Δεν πάει έτσι η εξίσωση αυτή είναι μια υποκειμενική ερμηνεία. Αντικειμενικώ δεν μπορεί να λέγεται αυτό. Υπάρχουν καταστάσει, πέραν των όσων υπόθηκαν, με στόλου που είναι πραγματικά απειρχιωμένοι. Εμεί όμω έχουμε και εφοπλιστέ που μα λένε ευχαρίστω να κάνουμε επενδύσει για να μειώσουμε τι δυνατότητε και τελικά δεν γίνεται τίποτα διότι συνεχίζει να υπάρχει, να, λειτουργεί ο ίδιος τόλος χωρίς εξυγχρονισμό και χωρίς να σταματάει και να περιορίζεται στις δυνατότητές του. Δεν γίνεται λοιπόν τίποτα έτσι, χρειάζονται επιδοτήσεις. Το κοινοβούλιο από τη Σκοπιά αυτή μου φάνηκε πολύ σοφό στην πρόταση που είχε κάνει για το Ταμείο της Αλίας και της Θαλάσσιας Ζωής και πρέπει να σταματήσουμε αυτή την προσέγγιση. Είναι εδώ και 20 χρόνια που δεν στέλνουμε χρηματοδοτήσεις στον τομέα της αλίας και για τον εξοχρονισμό της του στόλου. Περισσότερες επιδοτήσεις δεν σημαίνουν λοιπόν αναγκαστικά υπεραλίευση. Και μία ακόμη ερώτηση. Η μελέτη αυτή στρέφεται στα θέματα, το, στο θέμα των αλλιευμάτων και μας λέει η ε, μελέτη ότι είναι πολύ περίπλοκο να υπολογίσουμε την κατάσταση των αποθεμάτων. Ακόμη πιο περίπλοκο από ό,τι μα παρουσιάζεται εδώ, θα έλεγα εγώ. Διότι η πολιτική τη αλληλεία έπρεπε να έχει τρει διαστάσει. Περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική, οι οποίε είναι και δια, Αυτό δεν το λέει η μελέτη. Η προσέγγιση που έχει κατησχίσει τα τελευταία χρόνια, που έχει περισχύσει μάλλον τα τελευταία χρόνια και στην πολιτική τη αλληλεία, είναι να ε, δώσουμε την προτεραιότητα στο περιβαλλοντική διάσταση, ξεχνώντα τα άλλα εδώ λοιπόν πρέπει να μην ξεχνάμε δείκτε όπω την απασχόληση που δημιουργείται στο χώρο τη ε, Αλία, τη μέσο όρο ηλικία των Αλιαίων και του στόλου, την, ε, ε, το μέσο όρο κέρδου που παράγεται, το ΑΕΠ, το ότι υπάρχουν διαφορετικέ του στόλου, μερικοί είναι αριστεχνικοί, άλλοι είναι βιομηχανικοί. Είναι περίπλοκο το φαινόμενο, ακόμη περισσότερο από ό,τι μα παρουσιάστηκε εδώ μέσα αυτή τη μελέτη. Κύριε Μπιτό. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομος, διότι ήδη και προηγουμένως είπα πολλά, αλλά λίγο με ε, ενόχλησε αυτή η παρουσίαση διότι ο μόνος τρόπος που βρίσκουμε για να διαχειριστούμε τα πράγματα της θάλασσας, της αλίας, είναι να λέμε ότι δεν θα παίρνουν αρκετά οι ψαράδες, να περιορίσουμε τι πληρωμέ του. Γι' αυτό λοιπόν ξαναζήτησα το λόγο. Λίγο να το κοιτάξουμε αυτό. Ε, πρέπει να δούμε τις φιλοδοξίες που έχουμε στις θάλασσε και να δούμε και την ποιότητα των οικοσυστημάτων, ώστε οι πόροι, τα αποθέματα να μην είναι πλέον παράγοντα περιοριστικό. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να έχουμε φιλόδοξε πολιτικέ τη θάλασσε μεν, αλλά όχι μόνο την κοινή ελευθερική πολιτική. Και θα ε, ε, επαναλάβω αυτά που είπε και ο γειτονά μου. Ε, πρέπει να μην έχουμε μόνο κατά νου την περιβαλλοντική διάσταση τη θάλασσα. Πρέπει να είναι πολύ πιο σφαιρική η πολιτική μα προσέγγιση και να συμπεριλαμβάνει και τι κλιματικέ παραμέτρου και τι περιβαλλοντικέ, ε, πέραν των όσων προστάζει και επιτάσσει η κοινή ελευθερική πολιτική. Διότι οι ψαράδε ε, δεν μπορούν να είναι εμπλεγμένοι στα δίχτυα αυτή τη λογική. Πρέπει να αφήσουμε τα οικοσυστήματα να λειτουργήσουν και να τα διαχειριστούμε τα ηχθικά μα, ε, του ηχθικού πόρου με τον καλύτερο τρόπο, αλλά να επιτρέπουμε στους αλληλείς ε, να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την κατακαιρματισμένη προσέγγιση και όχι μια γενική επισκόπηση. Εάν έχουμε ένα ποιοτικό οικοσύστημα στη θάλασσα, δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για κατακαιρματισμό, για υπεραλίευση, για μείωση των ε, αλλιευμάτων και των όγκων. Πρέπει να προσέξουμε την πληρωμή ευρωπαϊκών πόρων, το τι γίνεται εν πλώ, το αν τα σκάφη είναι εξυγχρονισμένα, αν διαχειριζόμαστε σωστά τα αποθέματα και τέλος να έχουμε μια συνολική προσέγγιση ώστε να υπάρχει υπεύθυνη διαχείριση των αλληλευτικών πόρων. Και πέραν του να κοιτάζουμε το οικονομικό κέρδος, να σκεφτούμε ότι είναι ένα κοινό αγαθό για τις μελλοντικέ γενιές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μου φάνηκε λίγο απογοητευτικό ότι δεν, αναφέρεται δεν αναφέρομαστε ιδιαίτερα για την ISIS. Ε, διάβασα εγώ δύο γραμμές ερχόμενες εδώ ε, σχετικά με τις δυσκολίες ε, αξιοπιστίας ακρίβειας των δεδομένων ISIS για τα αποθέματα. Για την μέγιστη βιώσιμη απόδοση υπάρχει ένας τρόπος από ό,τι να έχουμε πιστοποίηση MSY, για να το πούμε έτσι. Η δική μου η απορία είναι πώς εξασφαλίζουμε ότι οι αλληλείς δεν θα αναγκάζονται να περνούν από το ένα είδος στο άλλο διότι η ISIS αποφάσισε ότι το MSY δεν είναι καλό για τα επόμενα έτη. Αυτό το είχαμε συζητήσει. Για ένα παράλληλο δηλαδή μοντέλο προς την ISIS. Αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε ξαφνικές ευνηδιαστικές λήψεις αποφάσεων. Επίσης νομίζω στην πέμπτη σελίδα που αναφερόμαστε στον κίνδυνο του εθνικισμού και αναφερόμενοι στα λαϊκιστικά κόμματα ε, το, το Brexit δεν είναι εθνικιστικό κόμμα εξ όσων γνωρίζω και δεν θα ήθελα και εμάς να μας συμπεριλαμβάνετε σε αυτό. Ε, κοιτάξτε, οι επιστήμονε απλώ αναφέρουν τι κάνουν τα ψάρια. Δεν είναι, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τα ψάρια, λέει ο πρόεδρο. κυρία Ουλρίσσα, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Τις εκτιμώ, τις σημειώνω και νομίζω ότι όλες ε, σχετίζονται με τον τετραγωνισμό του κύκλου, λέει η ομιλήτρια τι είναι βιώσιμο για το τάδε ή το δίνα για τα ψάρια, αφενός και για τους αλληλείς αφετέρου. Συζήτηση παλαιότατη και η απάντηση δεν είναι ποτέ είτε άσπρη είτε μαύρη. Μεταξύ της ε, ακραίας συντήρησης ε, από τη μία άκρη και της προστασίας, από της απόλυτης προστασίας της κοινωνικής των αλλιέων από την άλλη υπάρχει ένα πεδίο ενδιάμεσο επιλογών. Έχουμε μία τούρτα, έτσι θα πρέπει να το σκεφτούμε, που δεν έχει άπειρα πιτάκια. Ε, πρέπει να σκεφτούμε ποιο είναι το μέγεθός της και πώς μπορούμε να την εκμεταλλευόμαστε. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να αυξήσουμε το μέγεθος της πίτας. Όσο μεγαλύτερη είναι η πίτα, τόσο πιο παραγωγικό είναι το πεδίο, δηλαδή το περιβάλλον, και τόσο πιο είναι και για τους αλείς και για τα ψάρια λέει ο μιλήτρια. Και στα συμπεράσματά μου είχα ίσως ε, ε, κάπως σύντομα ε, συνοψίσει ότι χρειαζόμαστε μια προσέγγιση οικοσυστημική. Χρειαζόμαστε λοιπόν ανάκτηση της παραγωγικότητας των ηχθείων βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής τους, λέει η ομιλήτρια, πώς μπορεί δηλαδή ένα ψάρι να μεγαλώσει, να γίνει ενήλικας ως άτομο και μετά να το ψαρίσουμε και να το φάμε. Λέει η ομιλήτρια. Για την είσαις. και τα 50% των απαθεμάτων που υπεραλλιεύουμε κτλ. Βεβαίως και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα ISIS όλα αυτά συνελέγησαν σε μια έκθεση του ΣΕΣΤΕΠΕ, αλλά είναι οι ΆΙΣΕΣ που είναι η πηγή και αν θέλετε ο εγγυητής της αξιοπιστίας της επιστημονικής των δεδομένων αυτών. Ε, μπορεί να μην είχε σημειωθεί με σαφήνεια στην παρουσίασή μου, αλλά έτσι είναι. Επανέρχομαι τώρα στις ενισχύσεις και ίσως είναι το πιο αντιφατικό ζήτημα πράγματι βρισκόμαστε σε αυτήν την αντιπαράθεση μεταξύ βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης προσέγγισης να προστατεύσουμε τα αποθέματα ή τους αλληλείς. Όλες οι μελέτες όμως δείχνουν σαφώς ότι ένα νεότερο σκάφος είναι ισχυρότερο σκάφος. Δεν είναι μόνο η ασφάλεια που βελτιώνεται, αλλά είναι νέος κινητήρας που μπορεί να σύρει μεγαλύτερο εξοπλισμό και επομένως μπορεί να παγιδεύσει περισσότερα ψάρια ανά μία πορεία. Επομένως ο καθένας από τους αλληλείς επί τους σκάφου αυτούς μπορεί να αλλιεύσει περισσότερο και άρα η πίτα μειώνεται περισσότερο. Και σας το λέω αυτό για να σας δείξω πόσο δύσκολες είναι οι επιλογές μας. Άρα πόσους αλληλείς θέλουμε να διατηρήσουμε και τι αλλιευτική ικανότητα θέλουμε να έχουμε συνολικά αναχώρα και περιοχή. Στην Μεσόγειο έχουμε πολύ παλαιά σκάφη, έχουμε μικρού μεγέθους κατά μέσον όδο εξοπλισμό, Και βλέπαμε ότι σε κάθε σύγκριση ένα μεγαλύτερο σκαρί είχε μεγαλύτερη αλληλευτική δυνατότητα από τα μικρότερα. Με τάση Προ την υπεραλίευση, προς την δραστηριότητα την υπεραλιευτική μεσαιρείτε του σκάφους αυτού. Ένα νεότερο σκάφος ψαρεύει καλύτερα και άρα περισσότερο. Αυτό δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Βελτιώνοντα την ασφάλεια των επιβενόντων, δηλαδή των αλλαίων. Ο Μπεχτχόν σας το είπε νωρίτερα, πρέπει επίσης να διατηρούμε υπόψη μας ότι καθώς βελτιώνονται τα αποθέματα στην Ευρώπη, η κερδοφορία επίσης είχε βελτιωθεί, το είπε και ο συνάδελφος, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των στόλων στην Ευρώπη είναι κερδοφόρες. Κερδοφόροι, με συγχωρείτε. Δεν είμαστε στην καταστροφική κατάσταση οικονομικά που ήμασταν τα 10 προηγούμενα χρόνια. Και στην Μεσόγειο έχουμε στόλους που είναι κερδοφοροί γιατί έχουν καλύτερη ισορροπία επιτύχει μεταξύ αποθέματος και αλλιέων. Επομένως αυτή η ε, επίμονη, απεσιόδοξη προσέγγιση για τους αλληλείς που πεθαίνουν από την πείνα κτλ. δεν υποστηρίζεται από τα μεγέθη που δείχνουν ότι και τα αποθέματα βελτιώνονται και η κερδοφορία ακόμα και χωρίς ενισχύσεις των αλλιέων. Εγώ σας λέω λοιπόν προσοχή, υπάρχει κίνδυνος, αλλά και προσοχή, η κατάσταση δεν είναι τόσο κακή, τόσο απεσιόδοξη όσο μερικέ φορέ περιγράφεται. Τώρα, στην πρώτη ερώτηση για την υποχρέωση εκφορτώσεων και σας ευχαριστώ που τη θέσατε, διότι πρόκειται για ερωτήματα που σχεδόν δεν έχουν απάντηση. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, να αγνοούμε ότι έχουμε υψηλότατες ποσοστώσεις που αγγίζουν το 80% μερικές φορές εκφορτώσεων στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας στο πρόβλημα. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Πραγματικό πρόβλημα. Οι υποχρεώσεις εκφορτώσεων ήταν μια απόπειρα ε, βίαιη και ευνηδιαστική να βρεθεί μια λύση και η οποία μας οδήγησε στη σημερινή κατάσταση του τέλματος ε, και της ακαμψίας θα έλεγα πολύ δύσκολη κατάσταση ώστε να υλοποιείται, να εφαρμόζεται ομαλά πρόβλημα που δεν έχουμε καταφέρει να, επιλύσει, να επιλύσουμε μέχρι σήμερα το θέμα υπάρχει παντού, όχι μόνο στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, στην ε, Χιλή, στην Ασία, παντού. Και είχα αναφερθεί στο καρότο και το μαστίγιο, δηλαδή μεταξύ των κινήτρων και των υποχρεώσεων και πάλι εκεί πρέπει να βρούμε μια ε, χρηστή ισορροπία. Έχουμε όμως μπλοκαριστεί σε μια ε, διάταξη υποχρέωση εκφορτώσεων η οποία είναι εξαιρετικά καμψή, δεν αφήνει το περιθώριο στους τοπικού φορεί να κινηθούν δεν μπορούμε όμω να αμφισβητήσουμε, να αγνοήσουμε ότι είναι σημαντικό πρόβλημα. Η λύση που έχουμε σήμερα δεν είναι τέλεια, αλλά και εδώ θα ήταν λάθο απλώ να την καταργήσουμε και να επανέλθουμε στην προηγούμενη κατάσταση, γιατί είδαμε και εκείνη σε τι είχε οδηγήσει. Όλα αυτά τα ερωτήματα, τα ζητήματα δεν είναι εύκολα. Πράγματι, και υπάρχουν μια σειρά προκλήσεων για τα επόμενα χρόνια της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τα μέλη καλό είναι να γνωρίζουν ότι στις 12 Νοεμβρίου θα έχουμε ακρόαση για τις υποχρεώσεις εκφορτώσεων και έχουμε νέους προσκεκλημένους στις 3 για να μας εξηγήσουν οι ενδιαφερόμενοι πώς κάνουν τη δουλειά του και πώ αλλάζουν τα πράγματα από τη μία χρονιά στην άλλη και από την μία περίοδο την αλλιευτική στην επόμενη. Για να ακούμε και τα πρακτικά και όχι μόνο τα θεωρητικά. Ευχαριστούμε την καθηγήτρια και πάμε στην τρίτη παρουσίαση, την εξωτερική διάσταση. Ο κύριος... Over to you. Ο κύριος Αράντα. Buenas tardes. Eh, Καλησπέρα σα. Είμαι ο Μαρτίν Αράντα από το Τεχνολογικό Ίδρυμα Άστη στην Ισπανία και θα σας παρουσιάσω το τρίτο θέμα που είναι εξωτερική διάσταση της κοινή αλληλευτική πολιτικής. Παρόμοια δομή και η δική μου παρουσίαση. Θα ξεκινήσω δηλαδή μιλώντας εν συντομία για την εξωτερική διάσταση, τι είναι, μετά θα περάσω στις πρόσφατες εξελίξεις θα μιλήσω για τις μελλοντικέ προκλήσεις. Θα αναφερθώ σε κάποιες μελλοντικές περιπτώσεων στο πλαίσιο αυτή εξωτερικής δράσης, τέσσερις συγκεκριμένα και έπειτα θα περάσω στα συμπεράσματα και στις υποδείξεις, στις τάσεις. Γιατί υπάρχει εξωτερική διάσταση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Γιατί υπάρχει εξωτερική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζουμε πολύ καλά. Γιατί υπάρχει προτίμηση για τα ψάρια αισθητή υπάρχει μεγάλη προτίμηση το 1 τέταρτο των ψαριών που αλλιεύονται από τους αλληλευτικούς στόλους της Ευρώπης προέρχονται από εξωτερικά ύδατα. Το λέει και ιστορία. Έχουμε ηχθειότοπους σε μακρινά μέρη του κόσμου που ήταν ε, πηγή φοδιασμού σε ψάρια πολύ νωρίτερα από τη δημιουργία της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. στη στην Γη, Ατλαντικός, Κεντροανατολικός, εκεί αλλιεύουν επίσης Ευρωπαϊκή Στόλη, μεταξύ άλλων. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σκάφηνε 300 στην ε, αλία μεγάλων αποστάσεων. και αλλιεύουν στους βασικότερους εχθειότοπους του κόσμου. Συμμετέχει ενεργά η Ένωση σε έξι οργανώσεις για τον τόνο, στον Ατλαντικό, στον Ινδικό, στον Ανατολικό Ειρηνικό, το Δυτικό Ειρηνικό και σε όλα τα μήκη και, μήκη και πλάτη του Bluefin Tuna. Συμμετέχει επίσης Ένωση σε άλλες οργανώσεις περιφερειακές γύρω από την Αρκτική, Μεσόγειο, Ατλαντικό Βόρειο Ατλαντικό. Βορειοδυτικό και πιο πρόσφατα Νότιο Ειρηνικό. Όχι για τόνο αυτή τη φορά, άλλα είδη. Επίσης, υπάρχουν ε, συμφωνίες ε, βιώσιμης ε, αλίευσης, 7 για τον τόνο, 5 μεικτές πέραν των κτηνοδών και έχουμε και δύο συμφωνίες ε, με τα Φερόες και με την Ορβηγία. Στα γραφήματα εδώ βλέπετε εύγλωτα ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Είμαστε στην τέταρτη θέση σε ό,τι αφορά τα αλλιεύματα υπερβαίνουν τα 5 εκατομμύρια τα αλλιεύματα επίσης. Είναι μεγαλύτερη αγορά αλλιευτικών προϊόντων, με βάση τη μόφα μιλάμε για 30 δις. Αυτή είναι η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ ελκυστική αγορά. Πρώτα, αυτά τα 30 δις περιλαμβάνει εισαγωγές και εξαγωγές, κυρίως εισαγωγές όμως, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ψάρια που προέρχονται από άλλες περιοχές του κόσμου. Επειδή είδατε το πολύ ξεκάθαρο γράφημα πριν που λέει ότι είμαστε μια αλλιευτική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο, παγκόσμιο ελληνικού. ήθελα να σας κάνω και ένα άλλο σχόλιο επ' αυτού. Δεν μιλάμε μόνο για τον μεγάλο όγκα αλλιευμάτων, δεν είναι αυτό μόνο που μας δίνει ε, μια πρώτο καθετήρια θα έλεγα, αν δούμε την Ινδονησία ή την Ινδία και τα άλλα πλανεκτήματα. Παρόλα αυτά η Ένωση μπορεί να ηγηθεί στην διεθνή αλληλευτική διακυβέρνηση. Καταρχάς, πρώτον είδαμε, είναι μεγάλη αγορά αλληλευτικών προϊόντων. Έχει πολλά αλλιεύματα, μεγάλο ογκαλιευμάτων και επίσης δημοσία έχει εκφράσει την επιθυμία της να είναι ηγέτης στην Ινδία κυβέρνηση. Δεν μιλάει όμως και ποτέ πολιτική για ηγεσία στα αλληλευτικά, αλλά λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιτύχει το στόχο της ενίσχυσης ε, των δυνατοτήτων ε, των αλληλευτικών ε, οργανώσεων. Η άλλη διαφορά είναι το θεσμικό πλαίσιο που έχουμε σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Πολύ ισχυρό θεσμικό πλαίσιο αλληλευτικό βασίζεται στην κοινή αλληλευτική πολιτική και τον βασικό κανονισμό που αφιερώνει ένα ολόκληρο τμήμα στην εξωτερική διάσταση αλλά και άλλες νόμιμες πράξεις, νομικές πράξεις όπως είναι ο κανονισμός για τη διαχείριση εξωτερικών ε, στόλων Έχουμε τον κανονισμό για τον, την υπηρεσία ελέγχου που ελέγχει την αλία σε ξένα ύδατα εκτός ένωσης και έχουμε και άλλα νομικά μέσα. Όπως είναι ο κανονισμός για την παράνομη αλία και αυτό έχει εξωτερική διάσταση. Έχουμε και άλλα όμως εργαλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε επιστημονικά ε, εργαλεία, τεχνικά εργαλεία πολύ σημαντικά που και αυτά ε, κάνουν τη διαφορά σε σχέση με άλλες αλληλευτικές ε, υπερδυνάμεις. Έχουμε τη ΣΤΕΣΦ, την Επιστημονική Επιτροπή, τα ερευνητικά ιδρύματα των κρατών μελών που στηρίζουν τα κράτη-μέλη όταν αυτά συμμετέχουν στο δίκτυο περιφερειακών οργανώσεων, οργάνωση αλίας, Έχουμε το ISIS, e το Συμβούλιο Εξέρευνησης Διέρευνησης Αλίας, που και αυτό χωρίς να είναι ευρωπαϊκό, εκεί έχουμε συμμετοχή από επιστημονικά Ινστιτούτα των Κρατών Μελών. Επίσης έχουμε διάφορες αντιπροσωπείες και κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι διατίθεται κονδύλια συγκεκριμένα για την αλία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλία το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το, μάλλον το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το ΕΤΑ, που οργανώνει επεξακά προγράμματα σε διάφορες χώρες. Και έπειτα έχουμε και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το ΕΤΠΑ. Περιλαμβάνει περισσότερο όπως είναι η Μακρονησία, για παράδειγμα. Και εκεί η Μαδέρα, η Αζόρα, η και η Κανάρι, συμμετέχουν με προγράμματα. Μέχρι και το Κάπο Βέρντε, το πράσινο κροτίδι. Άρα έχει έρνωση τη δυνατότητα να ηγηθεί της διεθνούς αλληλευτικής διακυβέρνησης. Πρόσφατα λοιπόν, τι εξελίξεις είχαμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε κάποια μέτρα. Από την τελευταία μεταρρύθμιση και πριν ακόμα. Είχαμε συμφωνίες θερικής σχέσης στον τομέα της αλίας για τον εφοδιασμό των αλλιευτικών ε, στόλων σε άλλα ύδατα για την επιστηστική ασφάλεια. Αλλά τώρα πρόκειται για αλλιευτικές συμφωνίες βιώσιμες με άλλους στόχους και άλλες προτεραιότητες όπως είναι η ανάπτυξη της αλίας στα παράκτια κράτη που δίνουν πρόσβαση στη, στον Ευρωπαϊκό Στόλο. Έχουμε επίσης το κανονισμό για του Ευρωπαϊκούς στόλους που αλλιεύουν εκτός υδάτων Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο το μεγαλύτερο έλεγχο των ε, αλλιευτικών δραστηριοτήτων αυτών των στόλων και αυτό προηγείται της τελευταία μεταρρύθμιση της κοινή ελληνική πολιτική έχουμε τη δημιουργία του Γνωπτικού Συμβολίου για την ε, αλία σε ανοιχτά ύδατα, σε μεγάλε αποστάσεις. Δίνει τεχνική υποστήριξη, παρέχει τεχνικές συμβουλές αυτό ο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόσφατα τι είδαμε. Είδαμε ότι συμμετέχει, όπως είπαμε, στις, ε, ε, στις περιφερειακούς, περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλλιάς της πόδα αυτές. Έχουμε δράσεις ε, διαχείρισης, συντήρησης για να αντιμετωπιστούν οξέα προβλήματα, όπως είναι να αντιμετωπιστεί παράνομη, αδήλωτη, άναρχη αλεία, να μειωθεί η υπεραλίευση και να πάψουν να εφαρμόζονται αλλιευτικές πρακτικές καταστροφικές όπως είναι τα παρασυρώμενα απλάδια. Programas y proyectos que se realizan a nivel regional, como Η ε, τα, ε, τα οι πρακτικές ε, τα των πτυριγίων του Καρχαρία και για τη νέα ποιες είναι οι προκλήσεις ακόμα που δεν είναι νέες γιατί είναι προβλήματα παλαιότερα που θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε για πολύ χρόνο πλεονάζουσα αλληλευτική δραστηριότητα, παράνομη αλία σε πολλές περιοχές, μηχανισμοί κατανομής. Σε σπόδα όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για την ανάγκη κατανομής των αλληλευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών που είναι μέλη αυτών των οργανώσεων. Και μια άλλη σημαντική πρόκληση είναι μια πιο ολιστική προσέγγιση ώστε να λαμβάνονται υπόψη ε, τα περιβαλλοντικά και κοινωνικονομικά ζητήματα στη διαχείριση της αλίας. Επίσης, ξέρουμε ότι υπάρχουν θαλάσσιες περιοχές όπου δεν υπάρχουν α, περιφερειακές διαχείρισης αλίας, πόδων. Δεν υπάρχει μια αρχή δηλαδή για τη διαχείριση ή τη, τη συντήρηση. Αρκτική για παράδειγμα. Κεντροανατολικός Ατλαντικός. Επίσης έχουμε νέους πόρους που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον για τα βενθοπελαγικά είδη για παράδειγμα. Πρέπει να δούμε τι επίπεδα εκμετάλλευση μπορεί να υπάρχουν και ποια κατανομή των ε, κερδών μεταξύ των διαφόρων χωρών. Κάποιοι έχουν τεχνική οικονομική δυνατότητα, κάποιοι δεν έχουν. Πώ θα τα ε, ισορροπήσουμε όλα αυτά. Και υπάρχει και το θέμα τη κοινωνική βιωσιμότητα αλίας. ιδίω ό,τι αφορά τις ε, συνθήκες εργασίας των πληρωμάτων που ε, είναι πάνω σε πλοία ε, άλλων χωρών που πλέουν στα ανοιχτά ύδατα και μπορεί να τις θεωρήσει κανείς μέχρι και συνθήκες ε, δουλείας. Όλα αυτά τα επισημαίνουμε, ιδιω στη ΦΑΟ, από κοινού μάλλον με τη ΦΑΟ και με την, οργάνωση, την Διεθνή Οργάνωση εργασία και τον Αυτιλιακό Οργανισμό, πολλά μπορούν να γίνουν, είναι μεγάλη πρόκληση αυτή. Λοιπόν, τώρα, μελέτε περιπτώσεων. Συγγνώμη, κυρία Ράντα, θα είμαι άδικο μαζί σα, αλλά σα παρακαλούσα να επιταχύνετε λίγο. Να έχουμε τέσσερις ε, μελέτες περιπτώσεων για τον τόνο, ε, πόδα για τον τόνο, Δύο μεγάλες ομάδες ε, υπάρχουν, ε, ομάδες συμφερόντων, αν μπορώ να το πω έτσι, για την εφαρμογή των ε, μέσων διαχείρισης σε αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες. Τι γίνεται με την κατάψυξη των υπεραλλιευμένων αλλιευμάτων οι χώρες, οι παράκτες έχουν θεμητό δικαίωμα να αναπτύξουν την δραστηριότητά τους. Τα παρασυρώμενα ε, απλάδια είναι ένα πρόβλημα. Έχουμε αποκλειστικέ οικονομικέ ζώνε σε διάφορε χώρε και εκεί δεν ξέρουμε πώ μπορούμε να τα ορίσουμε αυτά. Επίση με Μαυριτανία, Σενεγάλη και Γινέα Μπισάου έχουμε συμφωνίε βιώσιμη Υπάρχει μεγάλη πίεση επίσης στον ευρωπαϊκό στόλο. Είναι πολύ περιορισμένο το νομικό πλαίσιο. Άλλοι στόλοι δεν το έχουν. Τα κράτη, τα παράκτη αυτά εδώ δεν έχουν τα τεχνικά και τα επιστημονικά μέσα και επίσης χρειάζεται διαφάνεια για τη χρήση των κονδυλίων που πολλές φορές πράγματι χρησιμοποιείται για δημιουργία ε, υποδομών. Τα είπα για τη διεθνή αλληλευτική διακυβέρνηση. Είναι φυσικός ηγέτης ε, για τη ε, διαχείριση ωκεανών και αλίας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πρωτοβουλίες και επίσης όλα αυτά τα προβλήματα που ανέφερα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Για το Brexit, το είναι τέταρτη μελέτη αναγνωρίζουμε και είναι τεκμηριωμένο ότι υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο επιστημονικό, τεχνική συνεργασίας, διαχείριση, πολύ στέρεο και είναι σημαντικό, πρέπει να διατηρηθεί. Η σχετική σταθερότητα ίσως πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε με τις ποσοστώσεις ε, να κατοπρίζεται καλύτερη κατάσταση και η κατανομή των ε, αποθεμάτων και επίσης μια μονομερής εκμετάλλευση δεν θα έχει θετική, θετικό αντίκτυπο ούτε για τον κλάδο ούτε για τα ψάρια. Λέμε λοιπόν στα συμπεράσματα ότι ένωσε σε καλή θέση για να από του ηγέτε στην ε, αλληλευτική διακυβέρνηση. Ένα άλλο συμπέρασμα είναι ότι χρειάζονται υποδομέ, δημιουργία υποδομών στι ε, παράκτε χώρε και χρειάζεται συνεργασία ε, μεταξύ των πόδα και άλλων φορέων για να μην μείνουν αυτές οι χώρες πίσω και πρέπει να υπάρξει συνέχιση της συνεργασίας ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του. Άλλη συστάση, να βελτιωθεί η θεσμική δυνατότητα ε, εκτός των ε, χώρων της Ένωσης, ιδίως ανεψόμενες χώρες, να υπάρξει παροχή ενισχύσεων σε χώρες που επιτρέπουν σε ευρωπαϊκά σκάφη να λύουν στα εδατά τους. Θέλουμε όμως να υπάρχει διαφάνεια για να ξέρουμε τι, πού, πόσο ε, ψαρεύουν η τρίτη στόλη για να υπάρχουν κοινοί κανόνες. Επίσης, συνεργασία, ιδίως όταν έχουμε κοινούς πόρους σε διμερές και διεθνές επίπεδο και τέλος καλύτερο συντονισμός μεταξύ των ε, διαφόρων δωρητών για τα κονδύλια για να μην υπάρχει επικάλυψη. Είτε με άλλους ε, δωρητές, είτε με διεθνείς τράπεζες, όπως Παγκόσμια Τράπεζα κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Ενθαρρυντικά αυτό μας είπατε. Διότι τονίσατε ποια πάνε καλύτερα αλλά το θέμα είναι και τι κάνουμε ε, ήδη καλύτερα από τους περισσότερους γύρω μας. Κυρία Αγγιλέρα. Eh, Να ευχαριστήσω για τη μελέτη αυτή για την εξωτερική διάσταση που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική για τον τομέα των αλλιευτικών στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε το δυναμικό του, γνωρίζουμε τα ισχυρά του σημεία, τα πλεονεκτήματά του, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Έχουμε ζήτηση για αλλευτικά προϊόντα που δεν απο... είμαστε ικανοί να απορροφήσουμε. Και το 40% της συνολικής κατανάλωσης γίνεται μέσω εισαγωγών από τρίτες χώρες. Υπάρχει σημαντική λοιπόν κατανάλωση ελευτικών προϊόντων που σχετίζεται άμεσα με αυτήν την εξωτερική διάσταση. Ε, εγώ βρίσκω πολύ εύστοχο το στοιχείο μεταξύ των συστάσεων ότι οι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υψηλές απαιτήσει σε θέματα διαφάνειας, προέλευσης, φυτογενομικά, βιωσιμότητα περιβαλλοντική και κοινωνική. Τα πρότυπα λοιπόν αυτά θα πρέπει να μπορέσουμε να τα διαβιβάσουμε, να τα μεταλαμπαδεύσουμε και σε άλλες χώρες και αγορές. Όταν λοιπόν ο Ευρωπαϊκός Στόλος αλλιεύει σε τρίτες χώρες μέσω συμφωνίας αλλιευτικής, έχει φέρει μαζί του, προβαίνει στην αλλιευτική του δραστηριότητα με όλα αυτά, συμμορφούμενος με όλα αυτά τα πρότυπα, σε αντίθεση με τους τόλους τρίτων χωρών που οδηγούν σε, μια, σε ένα μειονέκτημα ανταγωνιστικό εις βάρος μας. Επομένως αυτήν τη διαφάνεια πρέπει να την απαιτούμε και στην εξωτερική διάσταση από τους εταίρους μας. Και μερικές φορές εξ όσων εγώ γνωρίζω είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολο σε αυτές τις ε, αλλιευτικές συμφωνίες όπως μου δόθηκε η ευκαιρία να δώσω μια επίσκεψη στην ε, Γουινέα Μπισάου δεν είναι κανείς καθόλου βέβαιος ότι όλες αυτές οι τομεακές πτυχές πολιτικής φθάνει τα πλεονεκτήματα, δηλαδή πράγματι φθάνουν στον τομέα προς τον οποίο προσπαθούμε να στοχεύσουμε και να υποστηρίξουμε. Επομένως είναι σωστό να τονίζουμε την ε, διάσταση αυτή που πολύ συχνά την παραμελούμε κάπως αλλά είναι εξίσου σημαντικό τα δικά μας προτιμά να μπορούμε μέσω αυτών των αλληλευτικών συμφωνιών να τα διαβιβάσουμε και σε άλλες χώρες. Βελτιώνοντας και τις αλλιευτικές τους ζώνες και περιοχές, είτε τη δυνατότητά τους συνολικά γιατί μπορεί να είναι χώρες λιγότερο ισχυρές οικονομικά, ακόμα όμως και πολύ προηγμένες χώρες οι οποίες απλά δεν τηρούν τις βέλτιστες αλλιευτικές πρακτικές. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν πώς μπορούμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επηρεάσουμε τις συμφωνίες αυτές ώστε να προσθέσουμε αυτές τις απαιτήσει διαφάνειας να τηρούνται και από τις άλλες πλευρές από τους εμπορικούς μας εταίρους. Ε, Ο κύριος Άλλαρτ, ευχαριστώ για αυτό που μόλις είπε και η κυρία Αγγιλέρα. Πολύ μου άρεσε η διάσταση του Brexit που αναφέρθηκε μόνο μία φορά, αν καλά διάβασα. Το τι θα γίνει με το σκληρό Brexit χωρίς συμφωνία. Είναι όμως ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι το Brexit είναι μεν πρόβλημα, αλλά το Brexit χωρίς συμφωνία όχι. Κάτι που θέλω να ρωτήσω για όσους συνέταξαν αυτή τη μελέτη κυρίως. Μ' αρέσει πολύ η, μια παράγραφο στη σελίδα 104 που λέει για την ε, επίλυση μακροδιαφορών. Έχει άμεση σχέση με τον Brexit αυτό που θα συμβεί τους προσεχείς μήνες. Ή τη σχέση μας με την Ισλανδία που είναι μια πολύ σημαντική διάσταση εδώ. Θα έπρεπε ίσως κάτι να μπει και στα συμπεράσματα εδώ. Διότι θέλουμε μια συμφωνία πολυμερή. Δεν θέλουμε να συμπεριφερθεί κανείς όπως η Ισλανδία ε, σε αυτή τη φάση. Είναι σημαντικό να περάσει αυτό και θα ήθελα να αναφερθεί και στα συμπεράσματα. Θα συνέστηνα πρόεδρε να το συμπεριλάβουμε στην ημερήσια διάταξη πολύ σύντομα. Το θέμα της Ισλανδίας και πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όσα έχουν συμβεί σε αυτές τις μακροδιαφορές, την επίλυση μακροδιαφορών και πώς θα μπορούσαμε να δούμε μια σχέση συνεργασίας με την κυβέρνηση του ΕΒ στην περίπτωση του Brexit. Ε, ευχαριστούμε. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Καλό είναι να υπάρχει και κάτι θετικό για τον Brexit, ε, κύριε Άλλαρντ, αλλά και αυτό που πέρα για την Ισλανδία. Η Επιτροπή στην τελευταία συνεδρίαση, νομίζω, μας είχε πει και τον Οκτώβριο υπάρχει μια συνάντηση με την Ισλανδία, τις νήσους Φερόες και την Νορβηγία και τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ξανάρθει η Επιτροπή για να μας τα πει. Εάν τώρα μπορώ να επιστρέψω στους συμβούλους μας του προσκεκλημένους μας. Θέλετε να απαντήσετε σε κάτι από αυτά που ακούσατε. Μία απάντηση στην κυρία Αγγιλέρα. Πώς θα μπορούσαμε να εγγυηθούμε ότι και οι στόλοι τρίτων χωρών θα τηρούσαν αυτά τα πρότυπα στα πλαίσια αλληλευτικών συμφωνιών. Πώς θα μπορούσαμε να τους δώσουμε κίνητρα ώστε να τηρούν και αυτοί αντίστοιχες πρακτικές και αντίστοιχα πρότυπα. όπως εκείνα που τηρεί το δικό μας πολύ αυστηρό και πλήρε νομοθετικό πλαίσιο. Μιλούμε για κυρίαρχες χώρες που ε, ε, επιβάλλουν τις δικές τους διατάξεις, τις νομοθετικές, τους δικούς τους στόλους. Οι τελευταίες ε, περιπτώσεις αλληλευτικών συμφωνιών που είδαμε είχαν απλώς μια ρήτρα μη διάκρισης. Δηλαδή, ότι η χώρα θα πρέπει να επιβάλλει τις ίδιες ε, διατάξεις για τη δικού τους δικούς της στόλους και τους στόλους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά με την έλλειψη μια σειρά ε, στοιχείων εξοπλισμού προκειμένου να προβαίνουν σε ελέγχους που εξακριβώνουν την συμμόρφωση αυτή είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Υπάρχει η τομεακή ενίσχυση αλλά είναι αρκετά δύσκολο ζήτημα πριν να πει κανεί ώστε να έχουμε μια πραγματική, ένα πραγματικό έλεγχο της στήριξη αυτή. Όσο για την ε, αντιπαράθεση σχετικά με τη ρέγκα, λέει ο μιλητή και άλλα είδη τα οποία αλίευε η Ισλανδία με τρόπο πολύ μονομερή, είναι ένα παράδειγμα μονομερούς στάσης και το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει συνολικά τα αποθέματα όταν μια χώρα μονομερός επιβάλλει δικά της ε, τάκ, ε, αγνοώντας την υπόλοιπη ισορροπία της ζώνης. Μαζί με την Ορβηγία, τις, τις ε, νήσους Φαρόε και τα λοιπά. Ε, έχουμε μελέτες λοιπόν που μας δείχνουν σε ποιες περιοχές κινούνται τα αποθέματα ανάλογα με την ηλικία τους και επί τη βάση αυτών των ενδείξεων βασίζουμε τις συστάσεις μας των τάκ και ποσοστώσεων για το ποιο στόλος μπορεί να αλλιεύει πού, στα δικά του ύδατα ή στα γειτονικά κτλ. Είναι ένα συνολικό πλαίσιο δηλαδή που απαιτείται. Thank you very much. I... Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι βέβαιο ότι όλα τα μέλη τη Επιτροπή μα εκτιμούν αυτή τη διεξοδική μελέτη. Βεβαίω, είναι πολλή δουλειά που έχετε κάνει, αλλά είναι και πολλά τα σημεία που πρέπει να τα ξαναδούμε και να παρακολουθούμε πώ εξελίσσονται. Διότι ο κίνδυνο με τέτοιου είδου μελέτε είναι να μπουν στο χρονοτούλαπο και στο ράφι και να μην ξανασχοληθεί κανεί μαζί του. Όμω σε καθένα από τα τρία τμήματα υπήρχε τουλάχιστον και ένα κομμάτι με συστάσει στο τέλο. Η δική μου προσωπική συμβουλή προ τα μέλη τη Επιτροπή είναι όταν θα σας προσκαλέσουμε πάλι σε κανένα χρόνο να δούμε τα σημεία που θίξατε στο τέλος ως συστάσεις και να δούμε και τι πρόοδος έχει επιτελεστεί. Θα είναι ένα χρήσιμο πλαίσιο για τα επόμενα τρία χρόνια της δουλειάς μας λοιπόν. Και πάλι σας ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Α, καλλιέργεια. Εάν σωστά θυμάμαι, το 2011, όταν η κοινή αλληλευτική πολιτική κινήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκαινιάστηκε κιόλα, ε, ε, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονό ότι δεν φτάνουμε στο πλήρω δυναμικό μα στην ανάπτυξη τη αδοτοκαλλιέργεια. Το συζητήσαμε τότε διαμακρών. Η μεταρρύθμιση τη ε, ΚΑΠ θα μα έβαζε στη, στο σωστό δρόμο. Όμω παρά τον ενθουσιασμό που εκφράστηκε τότε, δεν κάναμε και μεγάλη πρόοδο έκτοτε. Ο κύριος Λάνεμαν νομίζω Σωστά το λέω. Λάνεμαν, παρακαλώ έχετε το λόγο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχω ετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση για να έχουμε και κάποια βάση για τη συζήτηση και μετά να τεθούν ερωτήσεις. Μας ζητήσατε να σας παρουσιάσουμε τι δυναμικό έχει για να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια. Και αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο για να επιτύχουμε και του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη και του ευρωπαϊκού στόχου τη επιστημιστική ασφάλεια, τη οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, τη ε, διατήρηση των αλληλεπτικών αποθεμάτων κ.ο.κ. Πρόσφατα, σε τομεί όπω οι κλιματικέ αλλαγέ, η κυκλική οικονομία, η πράσινη οικονομία και τα βιωσιμότερα διατροφικά συστήματα που απαιτούν και οι πολίτε. Εάν κοιτάξουμε την υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βάσει των τελευταίων οικονομικών μελετών που δημοσίευσε το 2018 Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά, οι επιδόσει είναι ω εξή. Ανακάμπτουν. Υπάρχει σταθερή, ακόμη και κάπω συγκρατημένη βελτίωση. Έχουμε 75.000 θέσει εργασία στην Ευρώπη, πολλέ φορέ σε λιγότερο αναπτυγμένε παράκτιε περιοχέ περιοχή τη Πέθρου και με πολύ ποικιλόμορφη ανάπτυξη ανάλογα με το κράτο μέλο, ε, τι ε, θαλάσσιε λεκάνε, τα είδη που καλλιεργούνται. αλλά πολλέ φορέ οι δυσκολίε που αντιμετωπίζει ο χώρο είναι κοινό σε όλου. Είναι κοινέ σε όλου. γι' αυτό λοιπόν μιλάμε για υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ένα χώρο. Ε, μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αν δούμε την παγκόσμια παρηγογή ε, τη υδατοκαλλιέργεια είναι ο πιο γοργά αναπτυσσόμενο ε, χώρος παραγωγής τροφίμων στον κόσμο. Τα μισά από τα θαλάσσια προϊόντα που καταναλώνονται στον κόσμο προέρχονται από την φωτοκαλλιέργεια και από τη θάλασσα. Και δεν μας εκπλήσει αυτό, διότι πώς αλλιώς θα μπορέσουμε να, να θρέψουμε τον παγκόσμιο πληθυσμό που διαρκώς αυξάνεται χωρίς να εξαντλήσουμε τα θαλάσσια αποθέματά μας. Έχουμε ε, πολλές φορές ε, πλου, σπάνιου πόρου που θα έπρεπε να εξαντλήσουμε στη γη και στη θάλασσα, αν έπρεπε να αντλήσουμε από κύλο μα τα τρόφιμα, είναι το καλλιέργεια μα προσφέρει μια εναλλακτική. Τα λέω πολύ γρήγορα. Ε, εάν δούμε την παγκόσμια παραγωγή ε, και τη θαλάσσια παραγωγή, βλέπετε και περίπου τα ίδια αποτελέσματα με την προηγούμενη διαφάνεια. Στα αριστερά. Στα δεξιά βλέπετε το θαλάσσιο είναι αυτό που προέρχονται από την αλία και τα κόκκινα από την υδατοκαλλιέργεια. Υπάρχει μείωση στην αλλιευσή και σταθεροποίηση στην υδατοκαλλιέργεια. Έχει γίνει σταθερή παραγωγή από την υδατοκαλλιέργεια και ο τομέα αυτό δεν έχει ε, αναπτυχθεί πολύ σε όγκο την τελευταία δεκαετία. Αναφέρατε το 2011, αλλά δεν έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα ε, Το μερίδιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην παγκόσμια υδατοκαλλιέργεια είναι 1,2% ω προ τον όγκο και 1,9% ω προ την αξία του τι παράγει η πρωτοκαλλιέργεια παγκοσμίω. Το μερίδιο έχει μειωθεί διότι έχει αυξηθεί και η παγκόσμια ε, παραγωγή. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το 60% των ε, θαλάσσιων κατανάλωση θαλάσσιων προϊόντων καλύπτεται από εισαγωγέ. Τα προϊόντα ε, τη υδατοκαλλιέργεια είναι 20% τη κατανάλωση και τα ψάρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο το 10% τη κατανάλωσή μα και των όσων βρίσκονται στι αγορέ μα. Η ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια είναι υψηλή αξία. Ε, συμμορφώνεται με υψηλά πρότυπα ποιότητα και ανθρώπινη καθώ και ζωική ε, υγεία, καθώ και τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Σε σύγκριση τουλάχιστον με τα εισαγόμενα προϊόντα. Η υδατοκαλλιέργεια μπορεί να συμβάλλει στο να πετύχουμε και άλλου πολιτικού στόχου, λόγω χάρη την ε, περιβαλλοντική προστασία ή την καταπολέμηση, την απαλλαγή από τον άνθρακα δεν είναι λίγο αυτό, αν λάβουμε υπόψη ότι τα ότι τα οστρακοειδή έχουν τη δυνατότητα να καθαρίζουν τα νερά στους ποταμούς ε, και επίσης να καταπολέμουν τον ευθοφυσμό, το ίδιο και με τα φύκια. Εάν δείτε άλλους τομείς στα αριστερά, Ε, βλέπετε την αξία και στα δεξιά την, τον όγκο. Το πορτοκαλί είναι τα ψάρια της θάλασσας, το κόκκινο είναι αυτά από τα γλυκά νερά, τα, εσωτερικά ύδατα και μετά έχουμε τα οστρακοειδή με γαλάζιο. Βλέπετε ότι και πάλι βέβαια τα ψάρια, τα θαλάσσια προϊόντα τη θάλασσα είναι τη μεγαλύτερη αξία. Τα οστρακοειδή είναι ακόμα χαμηλότερα, αν και σταθερά. Ω προ την παραγωγή, τα ψάρια τη θάλασσα έχουν ανέβει. Αν το δείτε ένα κράτος μέλος, ο τομέας επικεντρώνεται σε ορισμένα είδη μόνο και σε μερικές μόνο χώρες. Πέντε κράτη-μέλη έχουν 70% του συνολικού όγκου παραγωγής στην Ευρώπη των 28. Δεν είναι και πολλοί. Βέβαια βλέπω ότι δεν τα βλέπετε καλά από μακριά. Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα είναι οι πέντε ψηλότερε στήλε στον πίνακα. Και μετά βλέπετε ότι ακολουθούν οι και οι υπόλοιποι. Ως προς τον όγκο. Αν δούμε τα είδη. Εννέα είδη είναι περίπου το 90% του συνολικού μας, της συνολικής μας παραγωγής και του προπολογισμού. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν να διαφοροποιήσουμε την παραγωγή. Μετά θα δούμε τις μεθόδους παραγωγής καθώς και την καλλιέργεια νέων ειδών που είναι στο περιθώριο προς στιγμή. Από τα εννέα είδη έχουμε το σολομό του Ατλαντικού, την, το λαβράκι, τα οστρακοειδή, τα μύδια και ούτω καθεξής. Τι κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει της κοινή αλληλευτικής πολιτικής δεν έχουμε ε, αυστηρούς κανόνες γιατί η υδατοκαλλιέργεια πρέπει να ακολουθήσει πολλές ε, προδιαγραφές του περιβάλλοντος, της θαλάσσιας πολιτικής, την οδηγία πλαίσιο, την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, ε, για τα αποπτηνά και τα οικοτόπους τους, για την ζωική ευζοία, για την κυκλική οικονομία και το καθεξής. Πάντως, η κοινή ελευθερική πολιτική το 2013 βασίζεται σε στρατηγικέ γραμμέ για τη βιώσιμη ανάπτυξη τη στρατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ε, τρει αυτέ γραμμέ προβλέπουν μια εθελούσια διαδικασία για την ε, συνεργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα κράτη-μέλη για να προωθήσουμε την αεφορία και να αντιμετωπίσουμε τι κοινέ προκλήσει που ανέφερα και προηγουμένω. Οι κατατηρίε γραμμέ βασίζονται σε τέσσερι προτεραιότητε. Το να μειώσουμε το διοικητικό άχθο, ε, να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε νερά και σε συγκεκριμένου χώρου, να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και να αξιοποιήσουμε τα ανταγωνιστικά μα πλεονεκτήματα με ίσου όρου παιχνιδιού και ανταγωνισμού. Οι κατευθυντήριε γραμμέ είναι αυτέ που καθοδηγούν την πολιτική μα με την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, όπω είναι γνωστή, το βλέπετε και στο διάγραμμα. Ε, υποστηρίζεται αυτό με αιτήσει στρατηγικέ εκθέσει, προγράμματα κυρίω, σχέδια που καταρτίζουν τα κράτη-μέλη τα ίδια για την πολιτική του και αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλία. Επιχειρησιακά προγράμματα για τα κονδύλια που θα λάβουν ε, είναι αυτό που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη βάσει των εθνικών του προγραμμάτων με συλλογικό στόχο 25% σε όγκο ήταν όταν πρώτο ξεκίνησε αυτό. 1,2 δις ευρώ από το Ταμείο Θάλασσας και Αλίας τόσα έχουν δοθεί μέχρι τώρα μόνο για την υδατοκαλλιέργεια. Αυτά διατίθενται. Πρέπει να δούμε βέβαια πώς αδαπανήθηκαν, διότι ε, σιγά σιγά τα πάμε καλύτερα ω προ τα ποσοστά απορρόφησης. Ένα άλλο στοιχείο είναι τα έγγραφα καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το πώς να εφαρμοστούν λόγω χάρη κατευθυντήρες γραμμές από τα κράτη-μέλη, πώς να εφαρμόζουν την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, ε, πώς να διοδοτούν μια φάρμα υδατοκαλλιέργεια. Επιτά συνεργαζόμαστε συστηματικά με σεμινάρια τεχνογνωσίας με τα κράτη-μέλη, με ανταλλαγή καλών πρακτικών, με συμμετοχή στα προγράμματα ημέν των ΔΕ, με συμμετοχή ενδιαφερομένων και ένα από τα συμβουλευτικά συμβούλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά ακριβώς την υδατοκαλλιέργεια. Πέρσι ξεκινήσαμε μια ενδιάμεση αναθεώρηση της ανοιχτής συντονισμού για να δούμε πώς τα πάει η πολιτική μας. Σύντομα θα έχουμε και ένα υπηρεσιακό σημείωμα για τη, με τα πορίσματα αυτή τη ενδιάμεση αναθεώρηση. Τα προκαταρκτικά συμπεράσματα είναι ότι βάσει των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών είδαμε να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στην υδατοκαλλιέργεια από την πλευρά τη αγορά. Υπάρχει καλύτερη γνώση δηλαδή του τι συμβαίνει στην αγορά είδαμε αυτό να λειτουργεί στα πλαίσια του Ταμείου για τη Θάλασσα και την Αλία. Τα περισσότερα κάτι μέλη υιοθέτησαν μια στρατηγική για την υδατοκαλλιέργεια και βλέπουμε αν υπάρχει και καλύτερη επικέντρωση στην έρευνα για τα θέματα αυτά. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν ε, κάνει βήματα για να μειώσουν το διοικητικό άχθος. Και πολλοί έχουν πετύχει καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων εθνικών φορέων, των διοικητικών υπηρεσιών που ασχολούνται με το θέμα αυτό έχουν ευθυγραμμίσει και μειώσει τι διοικητικέ υποχρεώσει. Μερικοί θέλουν να δημιουργήσουν μια θηρίδα ή μονοπευθυντική για όποιον θέλει να ε, ε, ξεκινήσει μία φαρμαδατοκαλλιέργεια. Επιταχυμένη λοιπόν διαδικασία και κάποιε φορέ μπορεί να χρειαστούν και τρία χρόνια για να καταφέρει κάποιο να ξεκινήσει. Δεν έχουμε συγκεκριμένου αριθμού αυτή τη στιγμή για να δούμε ότι αυτές, αυτά τα διαστήματα αναμονή έχουν πραγματικά μειωθεί δραστικά, αλλά υπάρχουν πιθανότητε να βελτιωθούν τα πράγματα στο μέλλον. Και μετά υπάρχει και το θέμα τη θαλάσσια χωροταξία. Εδώ υπάρχουν βελτιώσει στο να ενσωματώσουμε και την ευρωτοκαλλιέργεια στο όλο πρόγραμμα. Τα πήγα πολύ γρήγορα. Επόμενα βήματα. Ίσως να έχετε δει και θα το δείτε και την επόμενη εβδομάδα με τις ακροάσεις των υποψήφιων επιτρόπων, ε, ο κύριος Βιργίνιους Σινκέβιτσιους έχει αναλάβει την αρμοδιότητα, το χαρτοφυλάκιο από την ε, προτινόμενη πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να συνεχίσει την στρατηγική για την πληθυστική ασφάλεια και παραγωγή τροφίμων. Γι' αυτό θα πρέπει να ξαναδούμε και τι στρατηγικές κατευθύνε γραμμέ για την πρωτοκαλλιέργεια του 2013. Εδώ αυτή η αναθεώρηση με την επικαιροποίηση έχει να κάνει και με τα διδάγματα που αντλήσαμε από το παρελθόν. Αλλά θα λάβουμε υπόψη και προσφατότερε εξελίξει για να δούμε πώ η θεατοκαλλιέργεια μπορεί να συμβάλλει γενικότερα στου στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε τι προβληματικέ επιδόσει του τομέα, θα δούμε την δυνατότητα προσαρμογή και αναχέτηση των ε, επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, όπου μπορεί κανεί δηλαδή να ε, ε, καλλιεργεί ψάρια ταυτόχρονα στις ίδιε θαλάσσιες λεκάνες ή να εκτρέφει ψάρια στις ίδιες θαλάσσιες λεκάνες και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα στο μέλλον. Και μετά μπορούμε να κάνουμε καλύτερα προγράμματα για την υδατοκαλλιέργεια. Ε, και Και εδώ βλέπουμε και το, την ομάδα της γαλάζιας ανάπτυξης. Η δατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας γοργά αναπτυσσόμενος τομέας. 250, 250 προγράμματα χρηματοδοτούμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προέκυψαν τα τελευταία δύο χρόνια. Καινοτόμα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από το LIFE, ή μέσω των εργαλείων στήριξη των μικρομεσαίων. Πολλέ νέε ιδέε κυκλοφορούν, αλλά πρέπει τα αποτελέσματα να τα εκμεταλλευτούμε καλύτερα και να διαδοθούν περισσότερο. Είναι μέρο τη πολιτική για τη γαλάζια οικονομία που έχει εγκρίνει πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τα νέα συστήματα παραγωγή. Αυτή είναι μια εικόνα από μία παράκτια μονάδα στην ε, Ζηλανδία η οποία παράγει Ε, η οποία παράγει συγκεκριμένα ε, ψάρια ε, με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να υπάρχουν εκπομπές στο περιβάλλον και τα οποία διοχετεύονται στην αγορά. Αυτό είναι ψάρια που προωθούνται στην αγορά του Λουξεμβούργου και είναι τοπική σχεδόν η παραγωγή. Πολύ κοντά στους καταναλωτές, τα εστιατόρια που τα παραγγέλνουν, είναι βιώσιμη η αλυσίδα. Υπάρχει και το λεγόμενο aquaponics, ο συνδυασμός καλλιέργειας με παραγωγή τροφίμων. Χρησιμοποιούμε τις εκπομπές από την εκτροφή ψαριών ως λίπασμα, ε, λιπαντική λικοπριά για να το πω έτσι, για, για την καλλιέργεια τροφίμων. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό από την άποψη της ε, κυκλικής οικονομίας για να ενσωμετωθούν όλα αυτά στην τροφική αλυσίδα ή την παραγωγή τροφίμων και να εκμεταλλευτούμε όλε τι δυνατότητες που προσφέρονται. Ένα ακόμα βήμα. Παρακάτω στην τροφική αλυσίδα είναι να δούμε τις δυνατότητες των θικών. Ο τόνος τα έχει φάει όλα που μπορούσε να φάει. Ίσως να παίρναμε την πρωτεΐνη απευθείας από τα φύκια. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα προγράμματα εδώ ως προς τις ζωοτροφές ή τα τρόφιμα. Πάντως, οι μονάδες υδατοκαλλιεργίας περιμένουν μήπως αρχίσουν να παράγονται μικροφύκια, ε, τα οποία θα ήταν μια εναλλακτική μορφή ε, σύντησης των ψαριών. Σε κάθε περίπτωση τα φύκια είναι πολύτιμο υλικό για βιομηχανική χρήση για παραγωγή οικολογικών προϊόντων και αν δεν αρχίσουμε να παράγουμε στην Ευρώπη θα χρειαστεί να τα εισάγουμε από αλλού όπου δεν ελέγχουμε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές ούτε και τις εκπομπές ε, από την παραγωγή τέτοιου είδους τροφίμων. Έχουμε ένα φόρουμ γαλάζιας οικονομίας με ε, ενδιαφερομένους που θα ετοιμάσουν ένα χάρτη πορείας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σκοπεύουμε να ε, εφαρμόσουμε τις συστάσεις τους. Ακροτελεύτια παρατήρηση. Εξίσου σημαντική. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την πρόσληψη από το κοινό. Δηλαδή πώς καταλαβαίνουν οι καταναλωτές εάν είναι καλύτερο να πάρουν ένα ψάρι που έχει εκτραφεί από ένα που το ψάρεψαν και να το φάνε. Είναι πολύ απλό αυτό. Εδώ βλέπετε ένα κινητό, μια κινητή σχολική τάξη που ταξιδεύει σε διάφορες περιοχές και με, εικονική, με εικονικά μέσα μπορεί να δείξει πώς ε, μοιάζει ένα ψάρι στη μια ή στην άλλη περίπτωση και να ενημερώσει καλύτερα τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Όποτε μιλάμε για την κοινή ελευθερική πολιτική στις μέρες μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνήθω μιλάει για την κερδοφορία τη επιχείρηση, το πώ μπορεί να βελτιωθεί η κερδοφορία. Δεν μιλήσατε καθόλου για το χρήμα, για το ποσό που μπορεί να ε, κομίσει κανεί. Είναι καλέ οι πιθανότητε. Τι γίνεται σε σύγκριση με τα ψάρια που αλλιεύει στη θάλασσα, Διότι εδώ βλέπω και μια τεράστια δυνατότητα εμπορική. Την έχουμε αξιοποιήσει Ναι, αλλά αν δείτε ποια είναι η αξία, το είπα κάπου. Να το. Ο σολεμός του Αθλητικού είναι 14% στον όγκο, αλλά 25% προς την αξία λόγου χάρη. Ή ας πούμε το λεγόμενο βασιλικό ψάρι από την ε, Ζηλανδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξειδικευτεί σε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα και τα έχει πάει πολύ καλά. Υπάρχει κόσμος δηλαδή που βγάζει πολλά από όλο αυτό. Και εδώ Πρέπει να πούμε ότι στο εμπορικό κομμάτι και το 2018 τα πήγαμε καλά. Ωραία. Η κυρία Τόμας έτσι πρώτα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να πω ότι η δατοκαλλιέργεια είναι πολύ σημαντική περιοχή και πρέπει να την ε, προσέχουμε ιδιαίτερα γιατί είναι από τους ε, πιο ταχαίως αυξανόμενους τομείς της ε, παραγωγής τροφίμων. 6 με 8% αυξάνεται κάθε χρόνο. Άνω των 85.000 είναι οι της απασχόλησης και λόγω της οικονομικής χρήσης των τελευταίων ετών ε, η υδατοκαλλιέργεια αυξάνεται ακόμα ταχύτερα. Και μαζί με την τροφική παραγωγή που είναι η πρώτη της στόχευση δεν πρέπει να ξεχνούμε και εναλλακτικέ παραγωγές που έχουν σχέση με τη χρήση των αποθυμάτων. Ε, στη χώρα μας ε, η υδατοκαλλιέργεια είναι πάρα πολύ ε, αυξανόμενο, επιταχυμένο αυξανόμενος τομέας Το 2018 η συνολική παραγωγή στο λαβράκι έφτασε σε πολύ υψηλό τονάζ, αλλά έχουμε πλέον ένα εμπόδιο για την περαιτέρω ε, αύξηση, ανάπτυξη του τομέα που είναι η τα θεσμικά εμπόδια ε, και η καθυστέρηση στι αδειοδοτήσει και στην πιστοποίηση. Χρειάζεται καλύτερο συντονισμό τοπικά και περιφερειακά, όπως και εθνικά, ε, και επίσης ε, δεν δημοσιεύονται αρκετά συχνά, ε, δεν υπάρχει πλήρης ενημέρωση σχετικά με, τις, με τα πλεονεκτήματα του τομέα, όπου ιδιαίτερα στις παράκτιες ζώνες δεν είναι ανταγωνιστικός προς τις, προς τις υπόλοιπες μορφές παραδοσιακής αλίας. Γιατί και αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη του τομέα αυτού. Ε, πρόεδρε, έχουμε επαναλάβει τη σημασία της υδατοκαλλιέργειας και περιβαλλοντικά, όχι μόνο οικονομικά και κοινωνικά, για τη βελτίωση των συνδικών ζωής της παρακτίας ζώνης, ε, την ε, επιστηστική ασφάλεια και την βελτίωση της ευμέρειας των πολιτών. Έχουμε στοιχεία του ΦΑΟ που μας λέει ότι ε, η υδατοκαλλιέργεια αυξάνεται ταχύτερα από τους υπόλοιπους ε, τομείς ε, της αλίας. Το 2016 είχαμε 5,8 παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης. Αλλά την ίδια στιγμή στην Ευρώπη είχαμε επιβράδυνση, τελμάτωση ακόμα και μείωση. Ο, ο, δέκατος παγκόσμιος παραγωγής είναι η Νορβηγία ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά χαμηλά στην παγκόσμια κλίμακα. Τώρα, ε, λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της, ε, των πλεονεκτημάτων της ε, κατανάλωσης θαλασσίων τροφίμων θα αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση για ε, αλλιευτικά προϊόντα ε, και ε, την ίδια στιγμή έχουμε μια αγορά που κυριαρχείται από τις εισαγωγέ. Η δική μας παραγωγή εδώ καλύπτει μόνο το 10% της δικής μας ζήτησης που σημαίνει ότι προσφεύγουμε σε προϊόντα εισαγόμενα από τρίτες χώρες. Για το μέλλον θεωρούμε ότι θα πρέπει να ανακτήσουμε ε, έδαφος έναντι των εισαγωγών. Και ίσως ε, στο μέλλον, ποιος ξέρει, να εγκαταλείψουμε και την κτηνοτροφία και την αλληλεία και να αφιερωθούμε όλοι εμείς ή τα εγγόνια μας τέλος πάντων ε, σε ειδικά αγροκτήματα υδατοκαλλιέργειας. οι στρατηγικές, οι μελλοντικέ της πολιτικής αυτής, ε, τα διοικητικά εμπόδια, το θεσμικά πλαίσια, η εδαφική ε, διαχείριση είναι ε, στοιχεία όλο και πιο σημαντικά. ακούσαμε την συνάδελφα από την Κροατία για το πώς βελτιώνεται η αγορά αυτή, η παραγωγή αυτή στη δική της χώρα, αλλά συνολικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουμε μια ασήμαντη παραγωγή σε παγκοσμίο επίπεδο. Ήθελα λοιπόν να κλείσω λέγοντας ότι στο Ταμείο της Αλίας είχαμε δώσει μια πολύ φιλόδοξη διάσταση στην υδατοκαλλιέργεια. Ο εισηγητής ήταν ο Γκαβριέλ Μάτο, όπως όλοι ξέρουν λέει ο μιλητής. Ε, και μάλιστα είχε αλλάξει και ο τίτλος του, ταμείου ώστε να συμπεριλάβει και την υδατοκαλλιέργεια ακριβώς. Ε, όλα αυτά τα στήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα ψήφισε ε, ε, για να έχουμε όχι μόνο προβλέψεις του προϋπολογισμού αλλά και ενισχύσεις και χορηγίες για τους δυνητικούς παραγωγούς. Επομένως υπάρχει συνείδηση της σημασίας Τη παραγωγή αυτή και νομίζω ότι στο επόμενο ταμείο θα πρέπει να και δημοσιονομικά να έχει την, την θέση που τους ανήκει, που τους αξίζει. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου λέγονται διάφορα. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο μελητής. Δεν κατάλαβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να σχολιάσω το εξής για την ε, ε, επιχείρηση Ζήλαντα, αν ακούσαμε καλά, ε, υπάρχει το εξή στοιχείο. στα πρώτα χρόνια της ύπαρξής της αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα. Χρειάστηκε να βρουν μια ισορροπία μεταξύ της ποιοτικής παραγωγής αλλιευτικών προϊόντων μια αντιμετώπιση διαφόρων ζωονόσων της ποιότητας του νερού κτλ Και η δεύτερη δυσκολία που αντιμετώπισε η εταιρεία αυτή ήταν ότι η αρχική πορεία αυτή τη startup είχε υποστεί και επικρίσεις από την ε, Κομισιόν, διότι της είπαν ότι δεν είχε σεβαστεί τους στόχους, ότι έπρεπε να επιστρέψει ενισχύσεις, ε, ε, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο της Αλληλείας. Δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι η γραφειοκρατική δομή ε, σχεδόν στραγγάλισε την επιχείρηση αυτή και βρήκαν άλλη χρηματοδότηση εναλλακτική. Δάλλος δεν θα τα έχει καταφέρει. Επομένως, ε, ξαναλέω, κινδυνέψαμε ε, συλλογικά να στραγγαλίσουμε αυτήν την επιχείρηση πριν καλά-καλά γεννηθεί. Ε, θα πρέπει λοιπόν οι διατάξει τη χρησιμοποίηση των πόρων των ταμείων αυτών ε, να είναι πιο ευέλικτε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Η κυρία Κόντε. Ε, πρόεδρε, η παραγωγή υδατοκαλλιέργεια υφίσταται ύφεση ε, ε, με σημαντικό αντίκτυπο επί της αγοράς εργασία και τη Ιταλική και τη Ευρωπαϊκή Αγορα. Μιλούμε για 85.000 ανθρώπους ε, που κυρίως εργάζονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ε, στην Ιταλία έχουμε περίπου 800 κέντρα, 800.000 τόνους το χρόνο νοπών προϊόντων, δηλαδή το 40% της ε, συνολικής εθνικής παραγωγής. Έχουμε προϊόντα υψηλότητα της ποιότητας με διασφάλιση εγγυήσεις ποιότητας, ελέγχους και με πολύ καλές ε, προοπτικές ανάπτυξης, ε, καθότι οι εισαγωγέ από τις τρίτες χώρες είναι 70% αυτή τη στιγμή. Η υδατοκαλλιέργεια είναι μεταξύ των τομέων με, την μεγαλύτερη, με το μεγαλύτερο δυναμικό βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας ε, θέσεων απασχόλησης. Αλλά αυτή, αυτά τα ταμεία της, Ευρω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι πιο ευκόλως προσβάσιμα από τις επιχειρήσεις για να επιτρέπουν τα καινοτόμα έργα να προχωρούν. Επίσης υπάρχουν κάποιες προβληματικές ε, υγειονομικών διατάξεων και χρήσης ε, χημικών ουσιών ε, που πρέπει να ελέγχονται καλύτερα. Πρέπει λοιπόν να παρέχονται πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την χρήση αντιβιωτικών στην υδατοκαλλιέργεια, με τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και για το οικοσύστημα, για το περιβάλλον. Μιλώ για την μικροβιακή αντοχή, όλη την αλυσίδα την διατροφική, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς χρησιμοποιώντας εναλλακτικέ ουσίες προς ε, τα αντιβιωτικά. Επίσης ε, θα πρέπει οι πόροι ε, να είναι βιώσιμοι, όλες, όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται να προέρχονται μάλλον από βιώσιμους πόρους και στις τροφές που χρησιμοποιούνται γιατί πολύ συχνά ο τομέας λόγω κάποιας έλλειψης διαφάνειας στις ε, αναθέσεις τις εξωτερικές ε, πάσχει από μια ε, έλλειψη διαφάνειας εγγύησης ως προς τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί για τα τρόφιμα, για τις τροφές. Αλλά μπορεί να συμβάλλει με επαρκείς ελέγχους και με επαρκείς εγγύησεις και επιστοποιητικά μπορεί να συμβάλλει εξαιρετικά στην εσωτερική παραγωγή μας και την εξυπηρέτηση της ε, ζήτησης εσωτερικά. Κύριε Σάλιβα, συμφωνώ με τον κύριο Μιγιάν Μον που είπε για τις επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στον κλάδο και διαρωτώ με μήπως χάσαμε το πλοίο ως Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ, γιατί δόθηκαν πολλά χρήματα στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας αν δείτε όμως κάποια από τα στοιχεία, αύξηση στον όγκο από το 7 και μετά δεν υπάρχει. Μόνο μια αύξηση στην αξία των προϊόντων που έχουν πολιθεί. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο λοιπόν λέει ότι έχουμε αύξηση της τάξης του 23% ενώ ταυτόχρονα είχαμε και ποσοστό πληθωρισμού της τάξης του 17%. τελικά η υποστήριξη στη βιομηχανία αυτή αποδίδει. Οι επιδοτήσεις εξασφαλίζουν την επιστική ασφάλεια και σε άλλους τομείς. Είναι καινοτόμο. Πολλά αυτά που γίνονται, πολλά από αυτά που γίνονται είναι καινοτόμα τελικά Ποια θα είναι η απόδοση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν απαντήσετε, λέει ο Πρόεδρος, πείτε μας και τι επιδοτήσεις ε, δίνει το Ταμείο. Ή αν θέλει κάποιος ε, να διαφοροποιήσει την παραγωγή του από το βόλιο κρέας, κάτι που δεν θα πού πάει. Πάει στην κοινή γεωργική πολιτική ή στο Ταμείο για την Αλία και τη Θάλασσα. Οι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Γκάτε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστώ την Κομισιόν για την έκθεση αυτή που είναι πολύ ενθαρρυντική ως ανάγνωσμα. Βλέπουμε έναν τομέα σε αύξηση. Τα βιώσιμα τρόφιμα άλλωστε είναι κάτι που όλοι επιθυμούμε. Τα στοιχεία λοιπόν είναι θετικά. Και το ότι εργάζονται 75.000 άνθρωποι σε αυτό το κλάδο και αυτό είναι σημαντικό για διάφορες χώρες. Ένα ερώτημα έχω προς την Κομισιόν, τέλο πάντων να επιστήσω την προσοχή της στο εξή. Ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Τι θα κάνει η Κομισιόν για να υπάρχει αυτό το ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Όταν έχουμε παραγωγούς τρίτων χωρών ε, που σαν τα πρώτα του στην Ένωση, υπάρχουν ε, άλλες φάρμες αυτοκαλλιέργειας που λειτουργούν και χρόνια με... Δεν είναι ισότιμο το πεδίο ανταγωνισμού. Ουσιαστικά θέλω να αναφερθώ σε πέστροφα από την Τουρκία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για τα στοιχεία που μας παρουσίασε για την δατοκαλλιέργεια. Τα καταλάβαμε ότι θέλετε να μα πλασάρετε, ε, άσε να μην το πω έτσι, θέλετε να προωθήσετε την ατοκαλλιέργεια, υπάρχουν προκλήσεις, η ποιότητα, η σημασία για την υγεία κτλ. Η αναρμόνιση της υποστήριξης ε, θέτει ένα θέμα. Ποια είδη θέλουμε να προωθήσουμε. Θέλω να προωθήσουμε κάποια άλλα δεν εκτρέφουμε όλα τα είδη και τα είδη που εκτρέφουμε δεν έχουν όλα τον ίδιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο ή την ίδια ε, εκπομπή θερμοκυπιακών αερίων, ε, πρωτεΐνες κτλ. Για τα μύδια, 100 φορές λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα ε, εκλείεται όταν τα εκτρέφουμε από άλλα ψάρια. Αντίστοιχα ισχύει και με την εκτροφή ζώων και την παραγωγή ζωικών πρωτεϊνών. Δηλαδή καλύτερα είναι να εκτρέφουμε ψάρια από τη ζώα σε ό,τι αφορά ε, τις εκπομπές ε, του θερμοκηπίου. Αλλά για να δείτε και την καντίνα ή το σπατόιστατρο των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Σολομός πρημοδοτείται τα μάλα Τουλάχιστον να τον εκτρέφουμε εδώ και όχι από αλλού. Καλύτερα να το μελετήσουμε, θα έλεγα. Από πού προέρχεται ο Σολομός. Αλλά πέρα τη πλάκα. Υπάρχουν κάποια σαρκοφόρα ψάρια. Από πού έρχονται. Και μήπως καταναλώνουν άλλες πρωτεΐνες και μήπως ε, έχουν κάποιο πρόβλημα με τη ε, σε εκπομπές θερμοκηπιακών και τι τρώνε αυτά τα ψάρια τέλος πάντων. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Okay, thank you very much. Um, Ευχαριστώ πολύ. Δεν καταλαβαίνω οι καλλιεργητές, οι μεγάλες εταιρείες κατοκαλλιέργειας. Μπορεί να έχουν εκμεταλλεύσεις για εκατοντάδες αγελάδες και έχουν να περάσουν από ελέγχους το ένα το άλλο και περιμένουμε τώρα να γίνουν επενδύσεις ξαφνικά στην εντατοκαλλιέργεια. Γιατί και παρόλα αυτά γίνεται, αλλά δεν προχωράει. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουμε εκτάρια επεκταρίων καλλιέργεια με το αντίστοιχο του πράσινου σε γαλάζιο. Στην Ισπανία μόνο βλέπουμε κάτι να συμβαίνει. Αυτό είναι το θέμα. Είναι θέμα των κρατών μελών. Και αυτό που μας νοιάζει είναι τι παραπάνω μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να το καλλιεργήσουμε. Και μετά και το θέμα της βιωσιμότητας, της εφορίας και το τι ε, ζωοτροφές δίνουμε στα ψάρια τι εγγύσει έχουμε ότι δημιουργούμε ένα πρόβλημα καινούριο ε, προσπαθώντας να λύσουμε ένα άλλο. Θα ζητήσω από την Επιτροπή να απαντήσει, αλλά αν κάποιο από του συναδέλφου θεωρεί ότι δεν απαντήθηκε η ερώτησή του, θα έχουμε χρόνο και για δευτερολογίε ή επερωτήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που κάνατε. Τα γνωρίζουμε και μερικές φορές έχουμε και εμείς τέτοιες υπαρξιακές αναζητήσεις. Σωστά ακούστηκε ότι όταν αξιολογούμε και θα αξιολογήσουμε το Ταμείο Θάλασσας και Αλίας για την τρέχουσα περίοδο, θα δούμε ότι δεν έχει πάει καλά. Τα μεγαλύτερα προβλήματα. Θα προσπαθήσω να τα θίξω όλα τα σημεία που ακούστηκαν. Βασικό θέμα ανεπαρκής διοικητική στήριξη. Ναι, γι' αυτό είπα ότι βλέπουμε κάποια κάποια μέλη να εγκρίνουν νέου κανόνε. Κάποια άλλα να ευθυγραμμίζουν διαδικασίε αν και ακόμα απομένει πρόοδο να γίνει. Εάν σα λέω ότι μια φάρμα καλλιέργεια χρειάζεται χρόνια για να πάρει μια άδεια, το η αξιολόγηση, το στατηγικό περιβάλλον, η αποδοχή από το κοινό είναι ένα θέμα η πρόσβαση σε συγκεκριμένο τόπο ε, για να δημιουργηθεί μια καλλιέργεια Μπορεί να υπάρχει και δίπλα μια παραλία και να μην θέλει ο κόσμο. Δεν θέλει κανεί μια καλλιέργεια ε, στην ε, δίπλα πόρτα. Υπάρχουν και πολλέ προκαταλήψει. Έχετε δει εικόνε από μονάδε αυτοκαλλιέργεια στη Χιλή, άλλε περιοχέ του κόσμου, με ντοκιμαντέρ από τον κόσμο. Μερικοί φοβούνται ότι θα γίνει κάτι ανάλογο δίπλα του ή τέλο πάντων εκεί που κάνουν μπάνιο. Ακόμη και αν αυτό δεν ισχύει. Για το φεγγαρόψαρο της Ιλανδίας, να πω ότι Βλέπουμε λοιπόν εδώ να έχει ξεκινήσει μια σειρά για τους ωκεανούς ε, με ντοκιμαντέρ. Ε, κάθε φορά έχει ένα διαφορετικό θέμα. Η τελευταία εκπομπή ήταν για τις γυναίκες στην Αλία. Τώρα έχουμε για την υδατοκαλλιέργεια. Αυτό το εργοστάσιο λοιπόν σας προσκαλώ να το κοιτάξετε το ανάλογο ντοκιμαντέρ γιατί έχει ενδιαφέρον. Ναι, για την γραφειοκρατία με κάθε νέα πρόταση για το Ταμείο Θάλασσας και ε, Αλίας προσπαθούμε να μειώσουμε το διοικητικό άχθος. Αυτή είναι η πρότασή μας, αλλά είναι και ο κανονισμός των ε, κοινών διατάξεων και με το κοινό γεωργικό ταμείο και με τα ταμεία συνοχής και το κοινωνικό. Προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε. Πάντως, η νέα πρόταση θα προσπαθεί να επιβάλλει λιγότερο διοικητικό άρθρο, αλλά μετά έχει τη διοικητική μηχανή των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ζητά τίποτα πίσω, αλλά στι κατοχώρε λόγου χάρη υπάρχει συγκεκριμένη αρχή που ασχολείται με την εκτέλεση του πολιτισμού νομικό πλαισίου στι κατοχώρε. Δεν του κατηγορώ, αλλά κάπου θα υπάρξει και γραφειοκρατία στην όλη εξέλιξη της διαδικασίας. Τώρα από το Ευρωκοινοβούλιο θέλουμε να υπάρχει και λογοδοσία για την ε, εκτέλεση των ποσών. και για τα αντιβιωτικά ή τα εμβόλια, την υγεία των ψαριών. Ε, εδώ Βλέπουμε σε διεθνές επίπεδο να υπάρχει εντατική δουλειά και σε συνεργασία και με το Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και την ανάλογη υπηρεσία του ΟΗΕ, το οποίο είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικό. Η υδατοκαλλιεργία δεν πρέπει να καταστεί στην παραδοσιακή αλεία, φυσικά. Συμφωνώ. Αλλά αν πάτε σε ένα εστιατόριο, στι Ιταλικέ ακτέ, οπουδήποτε, και ρωτήσετε από πού έρχεται αυτό το ψάρι, οι περισσότεροι θα σα πούν μάλλον στο 90% των περιπτώσεων. Από τη θάλασσα, από τη θάλασσα μόλις το πιάσαμε. Και αν μετά πάει κανείς και κάνει έλεγχο, έγινε μια γρήγορη μελέτη και 2,5% των ψαριών έρχονταν πραγματικά από τη θάλασσα. Τα υπόλοιπα ήταν όλα από εκτροφία. Ο σερβιτόρος δεν το λέει αυτό στον πελάτη, είναι θέμα αντίληψη και πρόσληψη από το κοινό. Αν ρωτήσετε στην κατίνα των εστιατορίων του Ευρωκοινοβουλίου από πού έρχεται το ψάρι, θα σα πούνε ναι, ναι, άγριο είναι. Από τη θάλασσα. Δύσκολα θα σας πούνε μυστικά, ε, ναι, είναι από εκτροφείο. Αν δείτε τι γίνεται με την υπεραλήψη στη Μεσόγειο, ίσως είναι καλό το 2,5%. Σε κάθε περίπτωση, πώς θα πετύχουμε να πάρουμε πίσω τα χρήματα που επενδύσαμε. Όταν αξιολογήσαμε το Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλία, κοιτάξαμε ακριβώς το πού και γιατί δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα. Δεν είναι το μόνο ταμείο που βλέπουμε άμεσα αποτελέσματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να το δούμε προσεκτικότερα. Ε, ρωτήσατε για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και την ε, αηφορία της τροφικής αλυσίδας το ανεφοδεσμένο στο τρόφιμα. Εάν δίνουμε ηχθιάλευρα ε, και ηχθιέλαια στα ψάρια εκτροφή, τι γίνεται με τα άλλα. Ναι, ναι, θα έρθω και σε αυτό. Πρώτα απ' όλα για τους ίσους κανόνες ανταγωνισμού. Και θα πω και για το δικό σας. Τι μπορούμε να κάνουμε με τους συναδέλφους μας στη Γενική Διεύθυνση Trade, το κοιτάμε, το γνωρίζουμε, Και όταν ε, υπάρχει τεκμηρίωση, λαμβάνουμε κατά ανάλογα μέτρα. Εξετάζουμε το θέμα και αν είναι θέμα θέμα του ανταγωνισμού, κοιτάζουμε ποια είναι τα αμυντικά μέσα που μπορούμε να εκδιπλώσουμε. Επίσης, ξεκινήσαμε και θα το ξέρετε, έχουμε και υγειονομικούς ελέγχους σε τρίτες χώρες κάποιες φορές και βλέπουμε πώς εκτρέφονται διαφορετικά είδη Ακόμα και βάσει των κανόνων του ΠΟΕ δεν μπορούμε να μπλοκάρουμε την πρόσβαση τέτοιων προϊόντων στις αγορές μας, αλλά πρέπει ο κόσμος να τα γνωρίζει. Ποια είδη είναι τα αγαπημένα μας και πώς τα εκτρέφουμε. Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να πάω σε μια νορβηγική μονάδα υφικαλλιέργειας Σολομών και οι Νορβηγοί μου λέγαν έχουμε κάνει σχεδόν φυτοφάγους τους Σολομούς μας. Εάν δείτε την εξέλιξη αυτή, εναλλακτικά τους δίνουν σόγια ή άλλα πρωτεϊνούχα τρόφιμα. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι χρειάζονται πόροι από αλλού. Γι' αυτό μίλησα για το Διεθνές Φόρουμ. Η Ευρωπαϊκή, ο Επίτροπος Βέλα είχε ζητήσει να λειτουργήσει ο μηχανισμός ε, Υψηλή υποπτία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πώ μπορούμε να, παίρουμε, να, να πάρουμε περισσότερου πόρου επιστημιστικού από του ωκεανού, ε, τα ταυτόχρονα τα αποθέματα. Δηλαδή, πρέπει να πάμε σε χαμηλότερα διατροφικά επίπεδα. Ε, πρέπει να εντοπίσουμε την πρωτενη στι αρχικέ τη πηγέ και όχι να περιμένουμε να φτάσει να έχει χωνευτεί επανειλημμένος, να έχει περάσει από τη διαδικασία της πέψης ξανά και ξανά για να τα δώσουμε στα ψάρια. Ένας τρόπος είναι να προσανατολίσουμε την γεωργία σε χαμηλής ε, πρωτεϊνικής ανάγκης ε, προϊόντα όπως τα οστρακοειδή, τα μαλάκια και άλλα που δεν είναι σαρκοφάγα αλλά φυτοφάγα. Να μια δυνατότητα ας πούμε. Και η άλλη εναλλακτική είναι να δούμε πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε την εκτροφή των ψαριών. Τα φύκια, τα φύκια μπορούν να καλλιεργηθούν και να αποτελέσουν αντικείμενα επεξεργασία με συγκεκριμένο τρόπο. Έχουν πολύ ψηλή θρεπτική αξία, περισσότερο από ότι τα ψάρια κάποιε φορέ. Ο Σολομό, λοιπόν, αν έχει χαμηλότερε ανάγκε, ε, εάν του δώσουμε ε, ζωοτροφή από φύκια, μπορεί να αυξήσει και την περιεκτικότητά του σε ω3 για τη χρηματοδότηση. Το 1, τα 1,2 δις που διατίθεται στον τομέα της θεατοκαλλιέργειας διανέμονται μεταξύ κρατών μελών. Τα, ε, τα, ε, τα ε, εκτελούν και τα εξοδεύουν, τα δαπανούν οι κρατικές αρχές. Σε πρώτη φάση κοιτάζουμε αν έχουν δαπανηθεί σωστά, αν έχουν μάλλον καν δαπανηθεί και μετά αν έχουν δαπανηθεί σωστά. Ο ετήσιος ρυθμός απορρόφησης είναι 50%. Κάτι λιγότερο από το 50%. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το ότι το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο ξεκίνησε σχετικά αργά. Αυτά προ στιγμή. Να λέμε στη διάθεσή σα για επιπλέον ερωτήσει. Uh, Υπάρχουν συμπληρωματικέ ερωτήσει. Μπιτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ μου φάνετε το λόγο à votre dernière intervention qui m'a un peu surpris. Je suis, je suis assez souvent d'accord avec vos prises de position. Δεν σας κρύβω πως εξεπλάγει ε, με την αναλογία που κάνατε εδώ, ότι θέλετε αυτές τις φάρμες ε, να τις παρομοιάσετε με μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ε, και αν δεν το ξέρετε σας λέω ότι είμαι Γιώργος και δεν καταλαβαίνω πώς δεν βλέπετε τι έγινε με τη γεωργική εκμετάλλευση, με τα πολύ παραγωγικά αυτά μοντέλα, τις μεγάλες αυτές δομές εκτροφής. 365 μέρες το χρόνο κλεισμένα τα ζώα χωρίς να φάνε ένα πράσινο φιλαράκι και να τα δει ο ήλιος και να τρώνε σόγια και καλαμπόκι ή χρήση μαζική γενετικώς τροποποιημένων, μεταλλαγμένων πολύ νερό επίσης ε, για την ε, παραγωγή και την καλλιέργεια σόγιας ε, και καλαμποκιού. Εδώ για το καλαμπόκι και στην άλλη πλευρά του για τη σόγια. Οπότε υπάρχει ένας φαύλος κύκλος με τέτοιου είδους ανάπτυξη εντό εισαγωγικών, ιδίω για την παραγωγή τροφίμων που σε ό,τι αφορά την ποιότητά τους καμία σχέση δεν έχουν, αν μείνω σε αυτή την αλογία, με τα φυτοφάγα που θα τρώγανε χορταράκι, ή το κρέας ή το γάλα αυτή, αυτά τα ζώα που είναι κλεισμένα ε, σε κλειστούς χώρους και τρώνε καλαμπόκι θα έχουν ε, αυτό που θα παράξουν ε, πλούσιο σε ωμέγα 6 λιπαρά. Αλλά τα ίδια ζώα σε ένα πιο παραδοσιακό και φυσικό περιβάλλον παράγουν μεν λιπαρά, ε, τρόφιμα πλούσια σε λιπαρά οξέα, αλλά όχι τα λιπαρά, ε, τα ω 6, αλλά τα ω 3, που είναι, δεν, είναι, δεν δημιουργούν φλεγμονές. Και on tire les enseignements de ce développement agricole de ces dernières décennies. Μην επαναλάβουμε τις λάθος αυτές πρακτικές ε, της τελευταίας δεκαετίας και στην υδατοκαλλιέργεια η ηχθειοκαλλιέργεια πλήττεται από τις λογικές που σήμερα λένε ότι θα επιτρέψουμε ε, να εισαγάγουμε το σολομό, γιατί μιλήσατε, για μεταλλαγμένο σολομό. Τι είναι ο μεταλλαγμένο ε, ε, σολομός με πολύ πιο γρήγορου ρυθμού ανάπτυξη, με αμφίβολης ποιότητας σάρκα, λόγω του αμφίβολης τροφής που, που παίρνει. Και πραγματικά σας χτυπάω το καμπανάκι και τα λέω φιλικά ε, απέναντι σας, γιατί συνήθως συμφωνώ μαζί σας, αλλά τώρα δεν. Συμφωνώ, με ανησυχεί κάπως η παρόμοιες που κάνατε, η αναλογία. Την έχω παρατηρήσει την ανάπτυξη Γιώργια, την τελευταία δεκαετία ή τις τελευταίες δεκαετίες. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος να βάλουμε στις ίδιες ράγες και την την υδατοκαλλιέργεια. Ξέρετε, εγώ δεν τρώω κρέας εδώ και 30 χρόνια, εν παρόδο. Ψάρια τρώω όμως, έτσι, μην ανησυχείτε. Απλά έλεγα, ε, είπα κάτι για την, αυτή την ε, παρομοίωση. Και στο Ρότερνταμ. χρησιμοποιούσαν ε, την ε, θερμότητα που περίσσευε από μια γειτονική ε, κατάσταση σε, κάποιο, σε κάποια εκμετάλλευση. Αυτό λέω. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ. Η υδατοκαλλιέργεια είπαμε ότι είναι ένας σημαντικός τομέας για την ευρωπαϊκή οικονομία και για την βιωσιμότητα του αλλιευτικού τομέα συνολικά ήδη αυτή τη στιγμή δίνει ε, δουλειά σε 85.000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός ο αριθμός αυξάνεται. Και μόνος καλά κάνουμε και ενισχύουμε την υδατοκαλλιέργεια, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε να μετατραπεί ένας ε, αλλιέας από τη μία μέρα στην άλλη σε υδατοκαλλιεργητή. Όπως είπατε και εσείς το 2% που, του ψαριού μόνο που καταλήγει στο τραπέζι μας προέρχεται από την παραδοσιακή αλληλεία. Αλλά ας ασχοληθούμε και με τους αλληλείς μια στιγμή. Ε, στη χώρα μας πολλοί αλληλείς θα ήθελαν να στραφούν στην υδατοκαλλιέργεια αλλά και να συμπληρώσουν την αλλιευτική τους παραδοσιακή δραστηριότητα αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρουν χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους γιατί η υδατοκαλλιέργεια απαιτεί επενδύσεις ε, σταθερές ε, προτού προλάβει κανείς να περάσει σε κερδοφόρα περίοδο η φάση, σε αντίθεση με την παρασιακή αλία και ε, απαιτείται και όλος αυτός ο γραφειοκρατικός οργανισμός, η δομή που συμπεριλαμβάνει τις περιφέρειες, το τοπικό επίπεδο κτλ. Ε, η Κομισιόν έχει κάποιο σχέδιο αντιμετώπισης ή ελάφρυνσης αυτού του γραφειοκρατικού ε, ε, μηχανισμού. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πλεονέκτημα σε κάποιες περιπτώσεις μετατροπής των αλλιέων ότι δεν τους πιάνει πια η θάλασσα, λέει ο πρόεδρος. Δεν, τους, δεν παθαίνουν πια ναυτία. Πολύ σύντομα. Um, δεν θέλω να παρέμβω στο πηγαδάκι σα εκεί, αλλά είπα ότι η αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών θα γίνει στο πλαίσιο τη πρωτοβουλία που ανήκει η πρόεδρο μελλοντική για τα βιώσιμα τρόφιμα και συστήματα. Δηλαδή θέλουμε βιωσιμότητα. Όχι στο επίπεδο του αγροκτήματο μόνο, αλλά και στο επίπεδο του πυρουνιού. Τι τρώμε δηλαδή και πώ φτάνει στο στόμα μα. From farm to fork. Δηλαδή τι σημαίνει από το αγρόκτημα μέχρι το πυρούν, μέχρι το πιάτο μας. Ε, αυτή είναι μια ολιστική προσέγγιση. Τώρα, κατευθυντήριες γραμμές θα αναθεωρηθούν βάσει και μιας ευρύτατης διαβούλευσης. Με την ίδια πάντα στρατηγική από το άγρισμα στο πιάτο και θα συζητήσουμε βέβαια και με τη δική σας επιτροπή τα στοιχεία που θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε σε αυτή τη νέα στρατηγική. Αν παρέχετε υποστήριξη για να περάσουν ε, ε, για να, γίνει, να υπάρξει περισσότερη ηχθιοκαλλιέργεια. Αλλαγή κατεύθυνση. Θα πρέπει να δούμε το τελικό σχέδιο, αν είναι δυνατόν. Αλλά δεν είναι στα χέρια της Κομισιόν. Στο πλαίσιο του νέου πολιτού, προσέγγιση που έχει προτιμηθεί είναι ότι ναι μεν θα δίνουμε δυνατότητα για περισσότερες επιλογές, θα καταγράψουμε όχι το τι θα στηρίζουμε, αλλά το τι δεν θα στηρίζουμε. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ αυτή την παρουσίαση. Το Κοινοβούλιο ανέκρινε μια έκθεση για την δατοκαλλιέργεια πριν από 15 μήνες περίπου. Μήπως είναι πρόωρο να ασχοληθούμε εκ νέου, αλλά είναι τεράστια ευκαιρία για τους Ευρωπαίους επιχειρηματίες με αυτός ο τομέας. Να περάσουμε στο τελευταίο σημείο, το υπαριθμόν 11, που είναι η διαδικασία απαλλαγή για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου της Αλίας. Με αυτή τη διαδικασία απαλλαγή μπορούμε να ασκήσουμε ένα εξονυχιστικό έλεγχο στο έργο του οργανισμού και αποφασίσαμε να συντάξουμε γνωμοδότηση την οποία και ανέλαβε η ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θα πάμε στον οργανισμό σε τρεις-τέσσερις εβδομάδες. Θα στείλουμε την προσωπία. Από την Κομισιόν, ποιος θα μας πει, αρενά, ή έτσι σας λένε. Ναι, καλησπέρα. Για την απαλλαγή τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου τη Αλία για το 2018. Επενούμε την υπηρεσία γιατί και το 2018 είχε ένα εξαιρετικό ποσοστό εκτέλεσης του προπολογισμού, στάξει το 99%. Η εφαρμογή και στις υποχρεώσεις και στις πληρωμές. 88 στις πληρωμές σε σχέση με το 74 της προηγούμενης χρονιάς και επαναλαμβάνω άλλη 99%. Η, το οικονομικό έτος αυτό, το 18, σημείωσε, σημειώ, σημαδεύεται από αυξημένες δραστηριότητες μετά από την πρωτοβουλία για τον πίνακα επιδόσεων ξεκίνησε το 2016 και ήταν η πρώτη χρονιά ενός project ε, στις ε, δικοαφρικανικές ε, χώρες για τη δημιουργία δυνατοτήτων. Παρά τις δυσκολίες που είχε η υπηρεσία, κατάφερε να διατηρήσει πολύ ικανοποιητικά επίπεδα εκτέλεσης του προπολογισμού και τις χαιρετίζουμε τις προσπάθειες αυτές. Επιβεβαιώνονται αυτά τα καλά αποτελέσματα και από την εσωτερική υπηρεσία ελέγχου της Κομισιόν. Πολύ θετική ήταν θετικό το πόρισμα του ελέγχου που έγινε το Σεπτέμβρη της περσινής χρονιάς. Σύμφωνα με το σχέδιο το στρατηγικό των εσωτερικών ελέγχων δεν εντοπίστηκαν κίνδυνοι, κρίσιμα σφάλματα σε ό,τι αφορά τον η ΕΦΚΑ είχε ήδη συντάξει ένα, σχέδιο δράσης για να μετριαστούν οι κίνδυνοι στο τομέα τη πληροφορικής. Κίνδυνος που εντοπίσει η εσωτερική υπηρεσία Ένα άλλο θέμα που πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το στάδιο και που είναι σημαντικό είναι ότι το Ευρωπαϊκό Λεγνητικό Συνέδριο για τη διαδικασία απαλλαγή του 2018 δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει την ετήσια έκθεση για τα αποτελέσματα των ετήσιων ε, λογιστικών ελέγχων των αποκεντρωμένων οργανισμών. Το περιμένουμε το έγγραφο αυτό με βάση τα αποτελέσματα των εκθέσεων που έχει εκπονήσει τα προηγούμενα χρόνια το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν πιστεύουμε, δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι θα αλλάξει η αξιολόγηση. Γιατί τα προηγούμενα έτη το ελεγκτικό συνέδριο έλεγε σε τελική γνώμη ότι υπήρχε νομιμότητα και κανονικότητα στην εκτέλεση των λογαριασμών. Τέλος. Ο οργανισμός εφάρμοσε όλα τα απαραίτητα μέτρα, έλαβε υπόψη όλες τι παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου και τι συστάσει από τη διαδικασία απαλλαγής του 2017. Δηλαδή, ήδη εφάρμοσαν όλα τα μέτρα σύμφωνα με το νέο χρηματοοικονομικό πλαίσιο 2018. Εδώ ολοκληρώνω την παρέμβασή μου και είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Λοιπόν, ίσως μπορεί να έχουμε ερωτήσει όταν επαστρέψουμε από την επίσκεψή μας στην υπηρεσία σας. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και με αυτό μπορώ να πάω στο 12, που είναι απλώς να σας πω ότι η συστάση των συντονισμών τον από την συνάντηση σήμερα το πρωί έχουν αποσταλεί με mail. Εάν δεν έχουμε σχόλια θα, θεωρηθώ, θα θεωρήσω ότι αυτά έχουν εγκριθεί. Εντάξει, ωραία. Δεν έχω κάτι, δεν μου έχει ζητηθεί κάτι από τα διάφορα. Και άρα, την ερχόμενη εβδομάδα θα ξανασυναντηθούμε, Τετάρτη στις 9